Good morning, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Έλεγχος των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. 23ος έλεγχος και πάλι σήμερα θα ξαναδούμε το IFMD και την Συμβουλή της ε, ΕΣΜΑ για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία και τους διαχειριστές αυτών. Και είχαμε συζητήσει την αρχική γνωμοδότηση της ε, ΕΣΜΑ για τα διαχειριστικά ταμεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε η γνωμοδότηση αφορούσε την εφαρμογή στο διοτήριο σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσι, Χονγκ Κόνγκ, Ελβετία, Σιγκαπούρη για την εφαρμογή της οδηγίας, κάτι το οποίο σήμαινε πως ε, η ανάλυση θα, μπορούσε, ε, θα αφορούσε μόνο μία συντομότερη περίοδο και άρα θα έπρεπε εν καιρό να ζητήσουμε ακόμη μία γνωμοδότηση για άλλες τρίτες χώρες και άρα είχαμε τον Ιούλιο του 2016 άλλη μία γνωμοδότηση που αφορούσε και αξιολόγηση χώρα μας ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσουμε τις λεπτομέρειες για την νέα αξιολόγηση της ΕΣΜΑ και την άποψη της Κομισιόν. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του IFNB, η Κομισιόν πρέπει να εγκρίνει μια πράξη κατεξουδότηση εντό τριών μηνών αφότου εκδώσει γνωμοδότηση η ΕΣΜΑ. Καλωσορίζω λοιπόν τους κυρίους Μέιτζορ και Γκέτνερ και έχετε τον λόγο για να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή. Παρακαλώ, Στίβεν. Uh, Ευχαριστώ, Ρομπέρτο, για την εισαγωγή. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ, αφού με προσκάλεσε ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΚΟ, να σας μιλήσω για τη δουλειά τη ΕΣΜΑ σε σχέση με το διαβατήριο στα πλαίσια τη οδηγία στις παρατηρήσεις μου θα συζητήσω την γνωμοδότηση για το κατά πώς θα πρέπει να επεκτείνουμε το διαβατήριο σε ξένες χώρες. Θα σας δώσω και κάποιες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα. Αλλά πριν περάσω στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης, θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή σε επετέχθη πολιτική συμφωνία για την οδηγία τον Οκτώβριο του 2010. Αντιμετωπίσαμε τη γνωμοδότηση για το αν θα επεκτείνουμε το διαβατήριο σε ξένες χώρες με απόλυτη προτεραιότητα και ξεκινήσαμε την προπαρασκευαστική δουλειά των στομπών των δυνατών. Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι αποφασίσαμε να αξιολογήσουμε τι ξένε χώρε μεμονωμένα και όχι ομαδικά. Το αποφασίσαμε αυτό γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ο μόνο τρόπο για να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση των διαφόρων κριτηρίων που καθορίζονται στην οδηγία. Ιδίω θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στι πολύ διαφορετικέ καταστάσει των ξένων χωρών σε ό,τι αφορά αυτούς τους παράγοντες ε, που αφορούν το διαβατήριο, την πρόσβαση ε, στις αγορές αυτών των ξένων χωρών για τα ευρωπαϊκά, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και διαχειριστές σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίζει η οδηγία. Αποφασίσαμε λοιπόν να εξετάσουμε μεμονωμένα την κάθε χώρα και εν συνεχεία να απτύξουμε μια πλήρη ε, μεθοδολογία αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια τη οδηγία. Δηλαδή, καταρχά, την προστασία των επενδυτών. Δεύτερον, την τι διαταραχέ στην αγορά. Τρίτον, τον ανταγωνισμό. Και τέταρτον και τελευταίο, την παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου. Η οδηγία προβλέπει ότι όταν η ΕΣΜΑ θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια για αυτά τα τέσσερα στοιχεία, η ΕΣΜΑ θα πρέπει να εκδώσει μια θετική γνωμοδότηση. Είναι σημαντικό να φέρουμε ότι η ΕΣΜΑ αξιολόγησε αυτές τις χώρες μόνο από κανονιστική και εποπτική σκοπιά και σας λέγουμε ότι άλλα θέματα, στην εκνομοδότησή μα, άλλα θέματα, όπω δημοσιονομικά θέματα ή θέματα κανόνων ξεπλήματο του χρήματο, που μπορεί να είναι σημαντικά για την απόφαση αν θα επεκτείνουμε το διαβατήριο, ε, δεν είναι δικά μα θέματα και δεν θεωρούμε ότι είμαστε αρμόδιο θέμα ε, σώμα να τα εξετάσει. Δημοσίευσαμε λοιπόν την πρώτη γνωμοδότηση τον Ιούλιο του 2015. Σε αυτή τη γνωμοδότηση αξιολογήσαμε έξι ξένε χώρε, το Γκέρνσι, το Χονγκ το Τζέρζι, την Ελβετία, τη Σιγκαπούρη και τι ΗΠΑ. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ο τέλειος τρόπος για να επιλέξουμε τις ε, ξένες χώρες, αλλά τις επιλέξαμε λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, το, λαμβάνοντας υπόψη και τις δραστηριότητες που έχουν οι οργανισμοί αυτών των χωρών υπό το Εθνικό Καθεστώς Ιδιωτικής Τοποθέτησης, NPPR. Ε, τη, γνώση και εμπειρία που έχουν οι δικές μας αρμόδιες εθνικές αρχές ε, απέναντι για τους ομολόγους τους η πρώτη γνωμοδότηση ήταν θετική για την ε, επέκταση του διαβατηρίου στο Γκέρνσι και στο Τζέρσι. Η Ελβετία επίσης αξιολογήθηκε θετικά. Θεωρήσαμε όμω ότι πρέπει να κάνει πρώτα κάποιε νομοθετικέ αλλαγές ε, για τις εξουσίες που έχουν οι εθνικές ε, ρυθμιστικέ αρχές. Και έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές. Αλλά δεν έχουμε πάρει τελική θέση για τι άλλε τρει χώρε. Σε αυτή την πρώτη γνωμοδότηση λέμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να αποφασίσουν να αναβάλουν την απόφαση για το αν θα ξεκινήσουν οι νομοθετικέ διαδικασίε μέχρι να, εκδώσει, μέχρι να εκδώσει ΕΣΜΑ θετική γνωμοδότηση για ένα μεγαλύτερο αριθμό ξένων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο θα λάβουμε υπόψη και άλλου παράγοντε όπω ε, την πιθανή επίπτωση στην αγορά για την απο, από την απόφαση να επεκτείνουμε το διαβατήριο. Το Δεκέμβριο του 2015 λάβαμε μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα ζήτησε να ερευνήσουμε επιπλέον δύο θέματα, κυρίως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κανόνων σε ξένες χώρες και μια προκαταρτική αξιολόγηση της αναμενόμενης εισρωής των οργανισμών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ξένες χώρες σε περίπτωση που το διαβατήριο επεκταθεί σε αυτές τις χώρες. Αυτή η επιστολή συμπεριλάμβανε και πλέον έξι ξένες χώρες που θα έπρεπε να αξιολογηθούν. Ε, η ΕΣΜΑ δημοσίευσε τη δεύτερη γνωμοδότηση για την επέκταση του διαβατηρίου στις 18 Ιουλίου του 2016. Σε αυτή τη δεύτερη γνωμοδότηση αξιολογήσαμε τις 12 ξένες χώρες συνολικά και λάβαμε υπόψη τις επιπλέον ανάγκες, τα επιπλέον αιτήματα που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή τη δεύτερη γνωμοδότηση ε, ήμασταν θετικοί για την επέκταση του διαβατηρίου στο Καναδά, Γκέρνσι, Χονγκ Ιαπωνία, Τζέρζι, Σιγκαπούρη και Ελβετία. Όμως, η ΕΣΜΑ σημείωσε ότι και το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη έχουν καθεστώτα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΟΣΕΚΑ μόνο κάποιων κρατών ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για μικροεπενδυτές στις επικρατείες τους. Για την Αυστραλία, η ΕΣΜΑ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια που να εμποδίσουν που να εμποδίζουν την εφαρμογή του διαβατηρίου υπό τον όρο ότι η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς της Αυστραλίας θα επεκτείνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ε, μαζικές ομαδικές αυτές εξαιρέσεις που αυτή τη στιγμή δίνει μόνο ε, σε κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με τις απαιτήσει ε, εφαρμογής του αυστραλέζικου κανονιστικού πλαισίου. Για τις ΗΠΑ η ΕΣΜΑ θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια για ταμεία τα οποία τα διαχειρίζονται οι διαχειριστές και απευθύνονται σε επαγγελματίε ε, επενδυτέ που δεν έχουν όμω δημόσια εγγραφή. Σε περίπτωση που υπάρχει όμω δημόσια εγγραφή, η πιθανή επέκταση του διαβατηρίου στι ΗΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ε, μη, συνθήκες μη ισότητας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι ε, θα έχουμε διαφορετικές συνθήκες ε, πρόσβασης στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στις Ηνωμένες και στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, για, τις δικές μας, για τους δικούς μας οργανισμούς οι οργανισμοί μας θα πρέπει να πληρώνουν πολύ περισσότερα. Επομένως, η ΕΣΜΑ θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν τι δυνατότητε για να μετριάσουν αυτού του κινδύνου. Για τη Βερμούδα και τα νησιά Κέιμαν δεν μπορέσαμε να αποφανθούμε οριστικά ε, για το θέμα τη προστασία των επενδυτών και την αποτελεσματικότητα τη εφαρμογή, μια και οι δύο χώρε είναι στη διαδικασία εφαρμογή νέων κανονιστικών καθεστώτων και η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη του τελικού κανόνε που θα ισχύουν στι δύο χώρε. Για το Isle of Man, η ΕΣΜΑ θεώρησε ότι η απουσία ενός αντίστοιχου καθεστώτος για μαθό της οδηγίας ε, ήταν καθεστώς δύσκολη την αξιολόγηση για το αν ε, η προστασία των επενδυτών ε, είναι παρκής. Ε, τώρα, μα, βραχυπρόθεσμα, θα συνεχίσουμε την αξιολόγηση της Βερμούδας και των νησιών Κέιμαν για να φτάσουμε σε οριστική, οριστικό συμπέρασμα το αν θα επεκτείνουμε το διαβατήριο σε αυτές τις χώρες. Δεύτερον, τι άλλο θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε την αξιολόγηση μιας τρίτης ομάδας ε, ξένων χωρών όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για τα επόμενα βήματα που σκέφτονται οι συνομοθέτε. Τρίτον, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα εκτεταμένο πλαίσιο, όπω αυτό προβλέπουν οι συνομοθέτε, σε περίπτωση που το διαβατήριο επεκταθεί σε μία ή περισσότερε ξένε χώρε. Αυτό το τελευταίο στοιχείο σημαίνει προετοιμασίε για το σημαντικό ρόλο που θα παίξει η ΕΣΜΑ για τη λειτουργία του διαβατηρίου και την ενίσχυση τη ε, εποπτική συνεργασία, που είναι προπόθεση για την επιτυχία. Θεωρώ ότι είμαστε στην κατάλληλη θέση για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, μια και θα βασιστούμε στην ε, δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, ε, προκειμένου να καταστήσουμε την, ε, τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές ανοιχτές σε οργανισμούς ξένων χωρών. Είμαι έτοιμος να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και ελπίζω να σας βοήθησαν αυτές τις αγωγικές μου παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Στίβεν. Ο Σβέν Γκέτνερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα στην Επιτροπή σας. Όταν συζητήσαμε την πρώτη ε, σύσταση της μας στην Επιτροπή σας εδώ, είχαμε τονίσει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες ε, των ε, χωρών και είχατε πει εσείς ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί και ο αντίκτυπος ε, των διαβατήρων σε τρίτες χώρες και το θέμα της φορολογίας και οι πτυχές ε, ξεβλήματος χρήματος. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν όλε αυτέ τι πτυχέ και το γεγονό ότι μόνο λίγε χώρε έχουν αξιολογηθεί, πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει μια νέα ε, προθεσμία για να υπάρχει μια πληρέστερη αξιολόγηση εκ μέρου τη ΕΣΜΟ που να καλύπτει περισσότερε χώρε. Όπω είπε ο Στίβεν, έγινε αυτό Συγκεκριμένα φέτος τον Ιούλιο στις 19 του μήνα λάβαμε εμείς την αξιολόγηση και τώρα αξιολογούμε αυτή τη σύσταση της ΕΣΜΑ. Τι μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα. Κατά την άποψή μας ε, η αξιολόγηση αυτή συνιστά σημαντική βελτίωση, ιδίω ό,τι αφορά την ε, επιβολή των κανόνων ε, για τη, οδηγίες για τους διαχειριστές σε τρίτες χώρες. Και βέβαια η ΕΣΜΑ έχει να αντιμετωπίσει μια πολύπλοκη πρόκληση σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία. Δύσκολα δηλαδή μπορεί κανείς να βρει δεδομένα, να βρει και τη σωστή μέθοδο για να δει αν μπορούσαν να υπάρξουν ε, διαταραχές και στρεβλώσεις ε, στην αγορά. Εξετάζουμε και κάποιες πτυχές ε, της εφαρμογής για να δούμε κατά πόσο μια τρίτη χώρα συγκεκριμένη θα μπορούσε να εξασφαλίσει και την εφαρμογή και την εποπτεία ώστε να εφαρμοστούν και να μην παρακάμπτονται οι κανόνε τη οδηγία. Θέλουμε να δούμε επίση αν οι εποπτικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βασιστούν εξ ολοκλήρου στου ρυθμιστέ των τρίτων χωρών για την εφαρμογή των κανόνων τη οδηγία. Τα μνημόνια συνεννόηση που έχουν συμφωνηθεί αποτελούν μια καλή βάση συνεργασία. Και ένα άλλο αν οι ρυθμιστέ των τρίτων χωρών θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ε, ευνίδιε αλλαγέ, ε, αλλαγή ποιων ε, κριτηρίων, τα και του διαχειριστέ κτλ. Όπω ήδη υπόθηκε, στην οδηγία απαιτείται από τι τρίτε χώρε να τηρήσουν τα πρότυπα της πρότυπης σύμβασης του ΟΣΑ. Ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ξεπλήματο χρήματο υπάρχουν αντίστοιχε διατάξει που πρέπει να τηρούνται από τι τρίτε χώρε. Επίση, τα κριτήρια για την στρέβλωση του ανταγωνισμού συνεπάγονται να δούμε παραμέτρου ό,τι αφορά το δίκαιο ανταγωνισμό. Όλε αυτέ οι πτυχέ δεν είχαν ενταχθεί στα καθήκοντα τη ΕΣΜΑ, άρα δεν αναφέρονται στη σύσταση. Και τώρα τα αξιολογούμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο αναλυτικά. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική καταπολέμηση τη φοροαποφυγή. Έχουμε πολλέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε για ενίσχυση τη συνεργασία εντό εσωτερική αγορά αλλά και με τι τρίτε χώρε. Προ τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα κατέθεσε ένα scoreboard, έναν πίνακα δικτών για τις τρίτες χώρες. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να οδηγήσει στην έγκριση του χρόνου ε, μιας λίστας για μη συνεργάσιμες τρίτες χώρες. Μεγάλα ο αριθμό των ζητημάτων που είναι ανοιχτά ακόμη. Δεν τα έχουμε αναλύσει απόλυτα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μα προ το παρόν ε, για το διαβατήριο στι τρίτε χώρε. Η χορήγηση διαβατήριου σε μια τρίτη χώρα δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι πολύπλοκο το περιβάλλον εντό του οποίου κινούμεθα, γι' αυτό και ακολουθούμε μια πολύ προσεκτική προσέγγιση. Θέλουμε να αξιολογήσουμε πλήρω εκτό τη ε, εισαγωγή του διαβατήριου. Δεν θέλουμε να διαστούμε στη λήψη απόφαση. Παροχή πληροφοριών για την αναμενόμενη έκβαση τη αξιολόγηση επίση είναι σε αυτό το στάδιο πρόορη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε μια πλήρη δέσμη κριτηρίων, την είδαμε τη δέσμη αυτή στο επίπεδο 1 και βασιζόμαστε και στα σχόλια που λαμβάνουμε και από τη δική σας Επιτροπή. Θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τις απόψεις των Ευρωβουλευτών για διάφορα ζητήματα τα οποία και προανέφερα. Και εδώ ολοκληρώνω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συμφωνώ και εγώ με την επιφυλακτική σας προσέγγιση. Λοιπόν, τώρα τον λόγο έχουν οι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα η συγγήτρια η κυρία Πιετικάινεν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους ε, της Επιτροπής αυτής ε, για αυτά τα οποία είπατε. Νομίζω πως η προσέγγιση που είχαμε ήταν μέχρι στιγμής στιβαρή και θα έλεγα πως ανταποκρίνεται στις αρχές μιας αρχής της προφύλαξης γιατί θα πρέπει σωστά να κάνουμε τα του διαβατηρίου. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, και μόλις άκουσα αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος για τα... Ο εκπρόσωπος Επιτροπής για τα σημεία αυτά της εξελόγησης. Ποιες πληροφορίες έχουμε, μπορούμε να βασιστούμε στην ικανότητα των τοπικών αρχών για την επίβλεψη, την επιβολή και τη συνεργασία. Δεύτερον, κάτι το οποίο συζητήθηκε αλλά δεν ήταν αντικείμενο της αξιολόγησης της ΕΣΜΑ αφορά τους κανόνες κατά του ξεπλήματος χρήματος και τα ζητήματα φορολογίας που έχουν όλο ένα και αυξανόμενη σημασία και σχετικό με αυτό είναι το ερώτημα πόσο χρόνο θεωρείτε ότι χρειάζεται μια αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών. Και το άλλο ερώτημα, τι θεωρείτε εσείς το κατάλληλο επίπεδο των χωρών αυτών για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού και επαρκείς πληροφορίες ε, για να κρίνουμε το πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, ε, οι κανόνες για να ισχύσει το διαβατήριο. Αν έχετε λοιπόν κάποια αξιολόγηση και μετά. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες γενικές κατευθύνσεις για το χρονοδιάγραμμα. Τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε. Όπως είπα, η δουλειά μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλή και καλό είναι να γίνουν ε, τα πράγματα σωστά και να γίνουν μία φορά από το να έχουμε μεμονωμένες βιαστικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Περβάνος Μπερέση για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ελίζα Φερέιρα παρακολουθεί το θέμα. εγώ τη σκητάλη τώρα εκ μέρου ε, τη ομάδα ω συντονίστρια. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΣΜΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι είναι σαν να βαδίζουν ε, πάνω σε αυγά. Τόσο προσεκτικά αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Ε, ακούσαμε τις δύο παρουσιάσεις και μπορούμε και εμείς να ζητήσουμε όλες αυτές τις ε, δυσκολίες που δείχνουν να προκύψουν σε σχέση με το διαβατήριο αυτό. Η νομοθεσία είναι επικριτική, όχι ότι επικρίνεται, είναι επικριτική και πρέπει και εμείς να είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των πιο δημιουργικών φορέων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον κύριο Μέιτσορ που ανέφερε το ζήτημα της φορολογίας και της καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος, το είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στη συνέχεια Φυσικά σε αυτό το τομέα για μας αυτό το σημείο έχει πολύ μεγάλη σημασία και ιδίω εν ώψη της τελικής αξιολόγησης για την δυνατότητα χωρίς αυτού του διαβατηρίου. Άρα δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση ε, προς το παρόν ε, ανεξαρτήτως της αξιολόγησης της ΕΣΜΑ όσο δηλαδή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουμε ε, επικύρωση σε θέματα φορολογίας δηλαδή ή ξεπλήματος χρήματος ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα δηλαδή. Όταν η ΕΣΜΑ μας λέει ότι για τις Βερμούδες και τις νήσους Κέιμαν ε, υπάρχουν προβλήματα και επειδή δεν είναι αυτοί που αξιολόγησαν ε, τις φορολογικές πτυχές ή τον κίνδυνο ξεπλήματος χρήματος, θα ήταν ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας να ακούσουμε ε, βασικά μέσω με ποια οπτική γωνία έχουν εκφράσει αυτές τις επιφυλάξεις και σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα για τη δυνατότητα εποπτείας. Έχουμε κάποιες ανησυχίες ε, ως προς αυτό το σημείο. Είπατε ότι δεν υπήρχε ισότιμη μεταχείριση των κρατών μελών, διότι ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αγορές του Χονγκ και της Σιγκαπούρης. Θα ήταν καλό να μας ε, αναπτύξετε περισσότερο το θέμα της ανισότητας αυτής, ανης μεταχείρισης. Επίσης, δύο θέματα θέλω να αναφέρω ακόμα. Πρώτον, πώς θα επηρεάσει αυτό το διαβατήριο τις ίδιες ευρωπαϊκές αγορές σε ποιο σημείο βρίσκεται η αξιολόγηση για τις χώρες για τις οποίες έχετε δεχθεί το διαβατήριο, για τους εσπέρους πάνω συνιστάτε να χορηγηθεί. Και ίσως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει βέβαια. Το επόμενο είναι ξεκινάμε και συνεχίζουμε την ε, μελέτη του θέματος, αλλά το διαρθρώνουμε με την ε, πιθανότατη κινητοποίηση το Μάρτιο του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί βλέπω ότι οι δύο πρώτες χώρες για τις οποίες δεν είχατε πρόβλημα ήταν το Γκέρζι και το Τζέρσι. Εδώ όμως έχουμε ένα πρόβλημα ε, που εξελίσσεται, μια δυναμική. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Thank you. Καμάλ. Ευχαριστώ, Σιέτ Καμάλ. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ΕΣΜΑ και την Κομισιόν. Ε, η ECR συζήτησε τα τελευταία χρόνια για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του διαβατηρίου και για την, την καθυστέρηση εφαρμογής ε, της οδηγίας, ε, την καθυστέρηση για την ε, ενσωμάτωση της οδηγίας ε, στην νομοθεσία των κρατών μελών, εμείς θέλουμε μια προσέγγιση αναχώρα και τις διακρίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές καταστάσεις σε ό,τι αφορά τη ζήτηση του διαβατηρίου, την πρόσβαση στις αγορές των οργανισμών και το νομοθετικό πλαίσιο στις τρίτες χώρες. Επίσης, με βάση το άρθρο 67 της οδηγίας, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δώσει θετική γνωμοδότηση ΕΣΜΑ για επαρκή αριθμό χωρών πριν ε, ξεκινήσουμε την νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται κυρίως στο άρθρο 65, 5 και 6. Το κριτήριο για την αξιολόγηση της οδυναμίας τρίτες χώρες υπάρχει στον πρώτο και έχει γίνει εκτεταμένη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ε, μας πήρε μήνες από τη ζωή μας, όσοι τουλάχιστον ασχοληθήκαμε. Και τα κάναμε όλα αυτά, ούτως ώστε οι τρίτες χώρες να έχουν καθεστώτα τα οποία προστατεύουν επαρκώς τους ε, καταναλωτές και μειώνουν τον κίνδυνο, το στιγμικό κίνδυνο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ε, αυτό σημαίνει και συνεργασία των αρμοδιών αρχών, προστασία των επενδυτών, ε, συμμόρφωση με τα άρθρα της οδηγίας, ε, διευθετήσεις για να μειωθούν οι, κινδύσεις, οι κίνδυνοι και ε, άσκηση των εποπτικών ε, εξουσιών από τις αρμόδιες ε, αρχές. η ευελιξία στην αξιολόγηση ε, υπάρχει στην αξιολόγηση που κάνουμε τις ΗΠΑ. Η ΕΣΜΑ θέλει θέλει να, εφαρμόσει το διαβατήριο σε δύο φάσεις. Επίσης, τι γίνεται με τα εθνικά καθεστώτα NPPR. Επίσης, θεωρώ ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να κάνουν θετική αξιολόγηση με βάση την, ε, τα όσα μας είπε η ΕΣΜΑ. Επίσης, η Κομισιόν ε, θα πρέπει να προχωρήσει αμελητή ε, για να χορηγήσει τα διαβατήρια σε τρίτες χώρες. Thank Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Τέσσερις ερωτήσεις έχω. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που περιμένει η Κομισιόν όσον αφορά την ε, επέκταση των διαβατηρίων για ένα περιορισμένο αριθμό τρίτων χωρών. Η Κομισιόν θα υιοθετήσει πράξεις κατεξιοδότηση σε αυτόν τον περιορισμένο αριθμό χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σκοπεύει να επεκτείνει περισσότερο τον κατάλογο τρίτων χωρών που θα λάβουν κάποια θετική απάντηση. Ποια είναι η προσέγγιση της Κομισιόν για τον σημαντικό στόχο και το διαβατήριο τρίτων χωρών θα δημιουργηθούν εταιρείες επένδυσης και ανάπτυξης για τους ε, Ευρωπαίους επενδυτές. Σε επιστολή του Δεκεμβρίου η Κομισιόν ζήτησε να, η ΕΣΜΑ ζήτησε να αξιολογηθεί πώς θα επηρεάσουν αυτά την εσωτερική αγορά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει η ΕΣΜΑ εάν έχει γίνει η μία τέτοια αξιολόγηση και αν ναι ποια είναι τα συμπεράσματα. Αν όχι, όταν ε, η ΕΣΜΑ θα επεκταθεί για να αξιολογήσει την ανταγωνιστικότητα των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων σε σχέση με τα καθεστώτα τρίτων χωρών. Πώς βλέπει η Κομισιόν το θέμα των διαβατηρίων σε τρίτες χώρες σε σχέση με το Brexit. Ας υποθέσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την ενιαία αγορά με αυτή την υπόθεση εργασίας πώς θεωρείτε ότι θα δοθεί το διαβατήριο τρίτης χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτομάτως θα δοθεί το διαβατήριο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση το γεγονός ότι συμμορφώνεται ήδη με τους κανόνες του EAFMD ή θα ακολουθήσετε μια άλλη προσέγγιση. Στο μέλλον, όσον αφορά τη χορήγηση αυτών των διαβατηρίων τρίτων χώρων, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι χώρες οι οποίες έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους κανόνες της ισοδυναμίας θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται και στο μέλλον και πώς θα έχει διαδικασία και ποιος θα την διοικεί. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Από την Όχι. Πράσινη λοιπόν. Δεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή, διότι για πολύ καιρό η Επιτροπή μας δεν είχε ουσιαστικά επεξεργαστεί τη χορήγηση διαβατηρίων και τα σχετικά, διότι μας έχει απασχολήσει πολύ περισσότερο η επικείμενη νομοθεσία. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δούμε πολύ πιο προσεκτικά τα ζητήματα της εφαρμογής και νομίζω ότι υπάρχουν δύο προφανή βασικά ζητήματα για τα οποία ισοτιμίες ή ε, τα διαβατήρια έχουν και μια πλέον πολιτική διάσταση. Πρώτον, οι στόχοι είναι πολύ πιο σοβαρή τη φορολογία και την ε, αντιμετώπιση του ξεπλήματος χρήματος αυτά τα δύο εργαλεία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση για τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει να είμαστε και αφελείς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια σαφή στρατηγική για τη χρήση των ε, σοδυνάμων αυτών και των διαβατηρίων. Ε, γιατί θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους καταπολέμησης των χρηματοοικονομικών εγκλημάτων. Δεύτερον, σημαντικό ζήτημα είναι το Brexit. Αν ακούσετε ή παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ε, Βρετανία. Σαΐτ, πολλοί συναδελφοί σου λένε ξεκάθαρα ας γίνει ένα έδος φορολογικού παραδείσου η Βρετανία, έτσι, στα ε, ε, περίχωρα, αν θέλεις, της ενιαίας αγορά Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ε, δεχθούμε, να δημιουργούνται όλο και περισσότερα προηγούμενα, δηλαδή τα οποία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα μα οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου θα έχουν χορηγηθεί αυτά τα εισοδήματα σε κάποιε χώρε από αυτέ τι συνθήκε και γιατί θα μα πούν δεν τα δίνετε στον καλύτερό σα φίλο που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί για να μην δημιουργήσουμε και άλλα προηγούμενα. Κανένας δεν θα πρέπει να πιστεύει ότι ένα προηγούμενο που δημιουργήθηκε στο παρελθόν τώρα μπορεί να συνεχιστεί να υφίσταται χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλες παράμετροι για το Ενωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν για το ζήτημα αυτό τη δημιουργία προηγουμένων, όπω είπε. Και κανεί δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο το ότι θα παραταθεί ε, ή θα επεκταθεί ε, λογικά η οποιαδήποτε χορήγηση διαβατηρίου σε αντίστοιχε συνθήκες. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα ε, σε ό,τι αφορά τη σύσταση. Ποια είναι η μεθοδολογία της ΕΣΜΑ για να καταλήξει αυτή τη σύσταση για την εφαρμογή της οδηγίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τα διαβατήρια στις τρίτες χώρες. Ε, μας ε, είπε ο Στίβεν ότι το 67-4 είναι η βάση. Αυτό το άρθρο ουσιαστικά αναφέρει την επενδυτική προστασία, διαταραχή της αγοράς, προστασία του ανταγωνισμού, παρακολούθηση συστημικών κινδύνων. Αυτά θεωρείται την βασική κίνδυνη στη δική σας, όμως καθοδήγηση η προσέγγιση ήταν πολύ πιο περιορισμένη, πιο περιοριστική. Επιλέξετε λίγα ζητήματα, αλλά δεν τα λάβατε υπόψη σε εκ τούτου, και συγκεκριμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν οι κανόνες που έχουμε για τη μόχλευση και τις αμοιβέ λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τα θέματα αυτά. Υπήρχαν επιθυμίες του Κοινοβουλίου, υπήρχε έντονη αντίσταση του Μεν Βασιλείου, αλλά ετέθησαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κάποιες θέσεις μας επεβίωσαν τελικά. Γιατί δεν λαμβάνονται λοιπόν τώρα υπόψη πλήρως αυτοί οι κανόνες για τη χορήξη του διαβατηρίου και τις οδύναμες αποφάσεις Και πιο αναλυτικά σας παρακαλώ να μας πείτε και οι δύο σας και από την ΕΣΜΑ και από την Κομισιόν. Τώρα, τι συνιστάτε, τι πρέπει να γίνει για να, είμαστε, να προχωρήσουμε σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων για την πρόσβαση στην ε, ενιαία αγορά μέσω του διαβατήριου. Πώς η Κομισιόν θα φτιάξει μια ευρύτερη και η ΕΣΜΑ πώς θα φροντίσει στις στάσεις της να λαμβάνονται υπόψη και τα ζητήματα που έχουμε, για το οποίο έχουμε αγωνιστεί εδώ και καιρό εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και εμείς. Το ENF ή το EFTT δεν εκπροσωπούνται εδώ βλέπω. Άρα, α, ναι, μπορούμε να δώσουμε τον λόγο πρώτα στην ΕΣΜΑ. Ε, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τα θετικά τους σχόλια. Να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ζητήματα που ακούστηκαν. Προτείνω τα ζητήματα φορολογίας να τα συζητήσει η Κομισιόν, γιατί όπως είπαμε η εντολή μας εστιάζεται στον κανονισμό και την εποπτεία και τα ζητήματα φορολογίας πρέπει να τα δούμε στον επόμενο γύρο όταν αποφασίσει η Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Επίσης νομίζω πως ως απάντηση στα σχόλια για το πώς λειτουργεί το σύστημα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το σύστημα το οποίο έχουμε εδώ με το FNB δεν είναι ένα σύστημα ισοδυναμίας. Σε ένα σύστημα ισοδυναμίας Μόλις μια χώρα θεωρηθεί ισοδύναμη, ουσιαστικά αποδέχεσαι όλη την εποπτεία, όλες τις ρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει άλλη πια εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό υπό αυτό το σύστημα, οπότε παρά τις αξιολογήσεις και παρά το ότι οι χώρες αυτές θα αξιολογηθούν και θα πάρουν το OK για το διαβατήριο, πρέπει να εγγραφούν ε, σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης και να συμμορφώνονται με τους κανόνες του AFMD. Οπότε για τα συγκεκριμένα ζητήματα της αμοιβή και της μόχλευσης θα υπάρχει ακόμα απέτηση για τους διαχειριστές των τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί στην Ένωση να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και να εφίστανται την εποπτεία. Οπότε δεν είναι ένα σύστημα ισοδυναμίας. Επίσης υπάρχει το μνημόνιο που πρέπει να συμφωνηθεί, το οποίο θα βοηθήσει τις ε, ρυθμιστικές αρχές, την Ένωση, έτσι ώστε οι διαχειριστές των τρίτων χωρών που θα εγγραφούν στην Ένωση θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του AFMD. Παραδείγματος χάρη, έχουμε απορρίψει κάποιες χώρες γιατί δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα μνημόνιο, γιατί δεν επέτρεπαν εξωτερικές επιθεωρήσεις για να δούμε αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ένωσης. Για τα πιο συγκεκριμένα σχόλια. του Χονγκ Κόνγκ και τα, κάποια οσέκα που έχουν προνομιούχο θέση εκεί πέρα και πολλούνται σε ε, επενδυτές λιανικής στο Χονγκ Κόνγκ και την προνομιακή θέση κάποιων κρατών μελών. Αυτό το λέμε γιατί υπάρχει κάτι το ασύνηθες από τις αρχές του Χονγκ Κόνγκ γιατί θα έλεγα πως έχουμε παρόμοια εποπτεία των ΟΣΕΚΑ στην Ένωση. Απ' την άλλη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το FNB ε, κατά βάση αφορά ε, επενδυτικά ταμεία λιανικής. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να πουληθούν σε τέτοιους επενδυτέ. και αυτή τη στιγμή είναι κάποιος, έχει το διαβατήριο, π.χ. ένα ταμείο του Χονγκ Κόνγκ που θα έρθει στην Ένωση, θα υπάρχει δυνατότητα ε, των κρατών μελών να εμποδίσουν την πώληση αυτών των προϊόντων σε καταναλωτές λιανικής. Ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το FNB κατά κύριο λόγο αφορά τα μία λιανικής. Για το θέμα των δύο στρώματων για τις ΙΠΑ, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν και γενικά υπάρχει μια λογική αμοιβαιότητα ή συγκρισιμότητα μεταξύ του να έρχονται εδώ αμερικανικά ταμεία και το αντίστροφο, εκτός αν υπάρχει βεβαίως μια εισαγωγή. Όταν υπάρχει εισαγωγή στο χρηματιστήριο, τότε φαίνεται πως είναι πιο δύσκολο για τα ευρωπαϊκά ταμεία να πάνε στη ΣΥΠΑ παρά το αντίστροφο. Οπότε, ένας τρόπος να το λάβουμε υπόψη είναι να επεκτείνουμε το διαβατήριο αυτό, όχι σε όλα τα ταμεία, τα επενδυτικά των ΗΠΑ, αλλά μόνο σε αυτά τα οποία δεν ε, κάνουν κάποιες εισαγωγές στο χρηματιστήριο ε, για το Brexit και τη συζήτηση τη σημερινή. Δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα έγινε ένα σχόλιο εάν θα υπάρξει μια ταυτόσιμη εφαρμογή. Πρέπει να δούμε βεβαίως τι θα επιλεγεί και εγώ ως τεχνικός δεν θα αναφερθώ σε αυτό, απλά να σε εξηγήσω τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες και το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Πράγματι, το FMD αφορά την εποπτεία, αλλά οι όροι της πρόσβασης δεν ορίζονται εκεί. Οι όροι της ε, πρόσβασης, τα ζητήματα της αμοιβαιότητα ε, δεν είναι κάτι το οποίο καθορίζεται στο FMD, είναι αυτό το οποίο συζητάμε εδώ σήμερα. Οπότε αν υπάρξει συζήτηση για αυτό το θέμα στο μέλλον, πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργούν οι διατάξεις περί πρόσβασης. Και επίση σχετικό για το Γκέρνσι και το Τζέρσι, κάναμε την αξιολόγηση σε αυτό το πλαίσιο με το, την τωρινή κατάσταση και την αντίληψη που έχουμε για τις δυνατότητες των ρυθμιστικών αρχών. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Τεχνική γιατί είπατε ότι η ΕΣΜΑ δεν χρειάζεται να δει ζητήματα ξεπλήματος χρήματος και φορολογίας. Απλά καλείται να δει ακριβώς ε, τα ζητήματα από πλευράς ε, εποπτείας της αγοράς το άρθρο 67 κτλ. Αλλά μετά το άρθρο λέει σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 35 και 37 έως 41 και στα άρθρα εκείνα γίνεται επίσης αναφορά σε φορολογικά ζητήματα και καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος. Ε, δεν σημαίνει λοιπόν αυτή η διάταξη ότι πρέπει να αξιολογήσετε και τα δύο κριτήρια, όχι μόνο τα τέσσερα που αναφέρονται, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία επιτρέπουν ε, στο διαβατήριο να λειτουργήσει σύμφωνα με τους κανόνες. Ε, καθαρά τεχνική νομική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, αυτά τα ζητήματα σχετίζονται ε, με τη φορολογία και αναφέρονται στο άρθρο το σχετικό που περιγράψατε. Πρόκειται για προαπαιτούμενο όμως. Υπογραφή δηλαδή ορισμένων εγγράφων. Τα ανέφερε ο εκπρόσωπο της Επιτροπής αυτά στην εισαγωγική του παρέμβαση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση άλλο το πραπετούμενο και άλλο τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 67 εδάφιο 4 το οποίο περιλαμβάνει τα κριτήρια για τον ανταγωνισμό. Εμείς αυτά τα κριτήρια εξολογήσαμε. Αυτό ήταν το πεδίο αρμοδιοτήτων και εντολή μας ε, ως ΕΣΜΑ. Οι φορολογικές πτυχές το ανταγωνισμό είναι κάτι που ε, πρέπει να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά και τον εκπρόσωπό τη. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις ε, για τον Brexit και τις επιπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να οικοτολογήσω εδώ για τα διάφορα σενάρια που αναφέρονται. Απλώς έχουμε μία πολύ προσεκτική και πλήρη προσέγγιση, λαμβάνουμε τα, τα πάντα υπόψη. Για να δώσουμε το διαβατήριο σε μια τρίτη χώρα απαιτεί λεπτομερή ανάλυση αυτή η απόφαση και χρειάζεται χρόνο φυσικά. Για τη συμμόρφωση των τρίτων χωρών ε, στα πλαίσια του διαβατηρίου και πώς θα λειτουργήσει. Εξαρτώμαστε από την ε, συνεργασία ε, των ε, εποπτικών αρχών μας και των εποπτικών αρχών των τρίτων χωρών με βάση το μνημόνιο συνεννόησης που έχει υπογραφεί. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να ανακαλέσουμε το διαβατήριο, αλλά ξέρετε πολύ καλά τι θα σήμαινε αυτό. Ακόμα και αν το δώσουμε. Σε ό,τι αφορά την φορολογία, εξετάζουμε όντως αυτά τα θέματα, το επιβεβαιώνω, το, ε, και είπαμε και στην εισαγωγική μας παρέμβαση, ότι εξαρτώμαστε από τη δουλειά που κάνουν σε διάφορα πεδία διάφοροι και εσείς εδώ στην Επιτροπή έχετε εξελίξει στον τομέα του ξεπλήματος χρήματος. Εμείς καταρτίζουμε στην Κομισιόν ένα κατάλογο. Αυτό συνδέεται και με το χρονοδιάγραμμα και με τα επόμενα βήματα. Εξαρτώμαθα λοιπόν από τη δουλειά που κάνουν σε άλλα φόρουμ, ούτως ώστε να έχουμε όλα τα στοιχεία για να πάρουμε απόφαση ε, για το διαβατήριο της τρίτες χώρες, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα φορολόγησης. Επιβεβαιώνω ότι εξετάζουμε το θέμα της ε, ισοδυναμίας και του διαβατηρίου από μια ευρύτερη σκοπιά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η κυρία Πιετικάνεν. Κανένας δεν σχολίασε το χρονοδιάγραμμα Θεωρείτε, πόσο χρόνο θεωρείτε θα μας πάρει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορείτε να σχολιάσετε τελικά και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Τα επόμενα βήματα. Η ΕΣΜΑ. Η Κομισιόν πρέπει να πει. Εμεί κάναμε ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που έπρεπε να κάνουμε, επομένως η Κομισιόν θα πρέπει να αποφασίσει τα επόμενα βήματα και πόσο χρόνο θα μας πάρουν. Όπως σας είπα, λέει η Κομισιόν, πρέπει να κάνουμε κάποια ανάλυση και εμείς σε ό,τι αφορά τα θέματα εφαρμογής των κανόνων και της ε, αποδιοργάνωσης της αγοράς. Και τι θα σήμαινε αυτό. Η δουλειά της ΕΣΜΑ έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει γίνει σε αυτά τα πεδία ε, και μας έχει δώσει τη γνωμοδότησή μας. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε πολύ προσεκτικοί, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν λαμβάνουμε απόφαση έχουμε όλα τα στοιχεία, όλους τους αποχρόντες λόγους. Και επίσης υπάρχουν και όλα τα θέματα των κειμένων τα οποία δεν εξαρτώνται. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα τα οποία εξετάζονται κτλ. δεν είναι στα χέρια μας όλα. Τα εξετάζουν άλλοι. Και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά σε άλλα, που γίνεται σε άλλα φόρουμ. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορώ να σας δώσω ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σημαντική ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων νομίζω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σωστά αυτά που είπε ο κύριος Γκέτνερ για τις επιπλέον επιπτώσεις που θα έχει η δουλειά που, που γίνεται και που δεν έχει τελειώσει ακόμα για θέματα φορολογικά και ξεπλήματος χρήματος. Likely acceptable by this committee to, to, to have a decision of passport which clearly would... Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δώσουμε διαβατήριο σε χώρες οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα σε, αυτά τα, σε αυτούς τους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν, για, θα έλεγα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις εξελίξεις και να δούμε ε, επίσης ποιες εξελίξεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας μας σε αυτά τα κρίσιμα παιδεία, σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς από τις χώρες αυτές. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, let's move to our points Οι συνάδελφοι περνάμε στα σημεία 9 και 10. Τίτλοποίηση. Όπως ξέρετε, στο τέλος Ιουλίου κατατέθηκαν γύρω στι 400 τροπολογίες για την πρόταση για το STS και άλλες τόσες για την πρόταση για το κοινού κανόνες ε, για την τυκλοποίηση και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ λύσεις. Κοινάμε λοιπόν από την απλή διαφανή, και, τυλο... και τυποποιημένη τυκλοποίηση. Ξεκινάμε τον Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό το κοινοβούλιο σε κάποια πράγματα στο ότι πρέπει όλοι να μάθουν τα διδάγματα της οικονομικής κρίσης και πρέπει να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή αν τα τοξικά προϊόντα πλέον δεν είναι τόσο τοξικά. Και το βάρος της αποδείξης βεβαίω το έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για να δώσουμε μια πιστική απάντηση εγώ περιμένω. Την στήριξη των συναδέλφων νομίζω μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πιστική απάντηση. Αλλιώς μια ισχνή πλειοψηφία θα γύρει αμφιβολίες και δεν θα είναι καλή αρχή. Λοιπόν, τεχνικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλουμε αγορές ε, βαθιές με ρευστότητα. Έτσι ώστε η να είναι μια αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης που χρειάζεται ε, να διαφοροποιήσει τον κίνδυνο από συστημικά σε μη συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να αποκαταστήσει και την εμπιστοσύνη στα τιτλοποιημένα προϊόντα για να μην αρχίσουν πάλι να τρέχουν οι επενδυτές σε καιρούς ασχημούς. Δεν είναι προφανές Βλέπουμε παραδείγματος χάρη δάνεια subprime για τα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ που δείχνει ότι και αυτή η αγορά πρέπει να οργανωθεί για να έχουμε ένα καλό προϊόν το οποίο θα είναι αντικείμενο εμπιστοσύνη. Για να έρθουμε τώρα στις ε, τροπολογίες ε, θα προσπαθήσω εγώ να ε, σας πω πού υπάρχουν οι δυνατότητες συμφωνίας αλλά και που υπάρχουν διαφωνίες. Μια πιο βαθιά αγορά με μεγαλύτερη ρευστότητα πρέπει να είναι διαφανής και πρέπει οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι υποπτικές αρχές να δουν ποια είναι τα διαθέσιμα προϊόντα και να έχουν πρόσβαση στα υποκείμενα δάνεια. Αλλά οι ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θέλουν να δουν αυτόν τον στόχο υπό τον όρο οι προτάσεις να είναι και ρεαλιστικές και αναλογικές. για να μην υπάρχει άλλη επικάλυψη προσπαθειών, αλλά να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά και ποια είναι τα στοιχεία, τα υποκείμενα των προϊόντων αυτών. Για τα συμφέροντα τώρα, νομίζω πως υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία πως η τιτλοποίηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα μοντέλο διασποράς της ε, πίστοσης, αλλά θα πρέπει ακριβώς να ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντά μας και πρέπει να το επιτύχουμε. Αυτό υπάρχουν πολλά στοιχεία στην πρόταση που απαιτούν περαιτέρω συζήτηση. Το ένα είναι το ποσοστό διακράτησης ε, του ρίσκου που έχουμε τροπολογίες που λένε να μείνει στο 5% μέχρι άλλες που λένε να φτάσει στο 25%. Οπότε τι το μέσο είναι γύρω στο 15%, αλλά βέβαια υπάρχει και η πιστοποίηση από τρίτα μέρη, Ποιο είναι υπεύθυνο και βεβαίω να δούμε και τι κυρώσει. Και θα πρέπει βεβαίως να συνδυάσουμε τα τρία αυτά σημεία. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί αλλά θα συζητηθεί είναι τα ABCP. Μια ομάδα θέλει να διαγραφούν εντελώς, αλλά κοιτούν την λήξη των δανείων, την μέση λήξη κτλ. Οπότε από τις διάφορες προτάσεις πρέπει να καταλέξουμε σε μία πάλι. Οπότε ε, δεν υπάρχει και χρόνος. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σκληρά για ναι, να βρούμε έναν συμβιβασμό με την ιδέα, όπως σας είπα, ότι χρειαζόμαστε αγορά με βάθος και ρευστότητα και θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αυτά τα προϊόντα κάνουν αυτό το οποίο υποτίθεται ότι κάνουν αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια πρόταση ε, συνεπή γιατί κάποιος μου είπε λύσατε τη μηχανή αλλά τώρα δεν είστε μηχανική και πρέπει να την ξανασυναρμολογήσετε. Αυτή είναι η δυσκολία. Για να έχουμε λοιπόν προϊόντα τίτλοποιημένα, απλά, διάφανη και τυποποιημένα πρέπει να έχουμε μια ε, σωστή πρόταση. Θα ακούσω λοιπόν τις προτάσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και ελπίζω οι πολιτικές ομάδες να σκεφτούν πώς θα επιτύχουμε μια συνεργαστική πρόταση με ε, πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Παύλος Θάλμπα ο εισηγητής της επόμενης έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η, αυτή η έκθεση και η επόμενη συνδέονται απόλυτα. Ε, συνεργάστηκα με τον Πολ και με τους υπόλοιπους ε, εισηγητές ε, και ευχαριστώ όχι μόνο τους κοιόδης εισηγητές αλλά και όλους τους αδέλφους που υπέβαλαν ε, τροπολογίες για να βελτιώσουμε τις δύο αυτές εκθέσεις. Ξέρουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αγορά τιτλοποίησης φυσικά είναι το πρώτο βήμα για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η αγορά τιτλοποίησης παίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας το έκανε πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης η τιτλοποίηση είχε λίγες ζημίες παρά το γεγονός ότι στιγματίστηκε κάτι που την επηρεάζει ακόμα. Επηρεάζει τη φήμη της αγοράς τιτλοποίησης και ακριβώς γι' αυτό συζητάμε σήμερα αυτές τις νέες προτάσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο στόχους να εξασφαλίσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και φυσικά να συνεισφέρουμε σε... και να εξασφαλίσουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω να εστιάσω στις ε, πιο σημαντικές πτυχές αυτής της έκθεσης. Καταρχάς, η ιεράρχηση των προσεγγίσεων. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν εισάγει διάφορες προτάσεις για το θέμα αυτό. Είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα αυτό της έκθεσης. Και θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθώ να βρω έναν τρόπο για να προσαρμόσουμε την ε, συμπερίληψη όλων αυτών των προσεγγίσεων και να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν τιμωρούνται όταν δημιουργούν INCs. Η Ένωση Κεφαλαίου Αγοράς, επίσης, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι μόνο για τους μεγάλους παίκτες. Ακριβώς το αντίθετο. Ότι θα πρέπει να είναι ένας διάβλος για να χρηματοδοτηθούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ευρύτατες επιλογές χρηματοδότησης και να μην βασίζονται μόνο στο τοπικό υποκατάστημά τους. Ε, θα πρέπει να έχουν διάφορες ε, δυνατότητες από επενδυτικά, επενδυτικές εταιρείες, από το leasing, από, από οπουδήποτε. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη δύο φορές, ε, με αυτά δηλαδή του παρελθόντος. Θα πρέπει να βάλουμε μπροστά στην ατζέντα, ψηλά στην ατζέντα της ημερήσιας της ε, μικρομεσαίας επιχειρήσης και είναι σημαντικό να συζητήσουμε δύο πράγματα. Για τη σύνθετη τυλοποίηση πώς θα υπάρξει ευελιξία ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία λύση που θα πρέπει να συζητήσουμε. Ε, Επίσης για τα ABCPs, για τα ιδιωτικά χρεογραφα καλυμμένα περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη οριμότητα, μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αλλιώς θα τιμωρήσουμε την δυνατότητα τυλοποίησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις κεφαλιακές απαιτήσει, νομίζω ότι η Κομισιόν ε, και το Συμβούλιο με τις προτάσεις τους πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση και φυσικά αυτό ε, συνδέεται με την υποχρέωση συγκράτησης του κινδύνου. Θα πρέπει να βρούμε μια συνολική λύση και για τα δύο θέματα. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που ήθελα να θέσω. Και περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας. Thank you very much. Ευχαριστώ. Äh, äh, Λέω meine Καταρχάς να ευχαριστήσω του δύο ε, και τους σκιώδει εισηγητέ, γιατί συνεργάστηκαν πολύ καλά. Αυτό που θέλουμε είναι η τιτλοποίηση να είναι ασφαλής τρόπος για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αυτό θέλουμε. Και υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο για πέντε άτομα, αλλά θέλουμε να δώσουμε ε, ζώνες για 7 άτομα θέλουμε να βάλουμε αερόσακους για 8 και μετά παραπονιόμαστε ότι το αυτοκίνητο δεν πάρει και τα γρήγορα. Ε, πρέπει να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν τεχνητοί φραγμοί. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι η τυλοποίηση είναι όλο και πιο ασφαλής και ότι έχει τις ε, επιθυμητές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε ασφάλεια και διαφάνεια. Παράλληλα, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι είναι και ελκυστική και ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε την τυπλοποίηση. Το να εξασφαλίσουμε και ασφάλεια και χρηστικότητα, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτή την ισορροπία, τη λεπτή ισορροπία δεν την έχουμε ακόμα βρει. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτή τη λεπτή ισορροπία, ούτω ώστε να υπάρξει ευρύτατη συνένεση. Καταρχά, ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Το αποθετήριο δεδομένων τυπλοποίηση. Ε, κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση με τους τρεις ε, φορείς που επιτρέπει η ΕΣΜΑ ε, θα μας εξασφαλίσουν επαρκή πραγματογνωμοσύνη. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει το κομμάτι αυτό. Για την ασφαλή τρίτη χώρα τώρα. Ή το καθεστώς της τρίτης χώρας ως προς την τίτλοποίηση, εκεί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν και δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα του STS χωρίς να αποκλείουμε κάποια τίτλοποίηση και βεβαίω να υπάρχει μια, ένας διαχωρισμός παλαιών και νέων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι παλαιές τιτλοποιήσεις ε, είναι άσχημες ή ότι φταίνε όλες οι φυστάμενες τιτλοποιήσεις για την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Η τρίτη πτυχή και παραμένει νομίζω ε, ως το βασικό πρόβλημα και θα κρίνει την επιτυχία της πρότασης είναι το 5% διακράτηση ρίσκου Κοιτάξτε, εγώ ξεκινάω με βάση πως αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν ε, στην ε, οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων 2 που έκρινε ότι το 5% είναι επαρκές και εξηγεί γιατί. Και βεβαίως και στην ΣΕΠΣ ε, ο Ευρωπαίος δηλαδή επόπτης το επιβεβαιώνει και η ΕΠΑ επίσης. Οπότε αυτή τη στιγμή Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να πάμε από το 5% στο 25% και ταυτόχρονα να παραμείνουν ελκυστικές οι τιτλοποιήσεις και να συμφωνήσουμε. Δεν είναι θέμα συμβιβασμού όταν είμαστε μεταξύ 5 και 25 να πούμε 15 γιατί το αποφασιστικό είναι η τιτλοποίηση. Ή να αυξήσουμε την ε, ελκυστικότητα, να αυξήσουμε την ασφάλεια χωρίς ε, βεβαίως αυτό να οδηγήσει σε αφανισμό αυτού του μέσου. Γι' αυτό δεν είμαι πεπισμένος ε, για το ότι πρέπει να φύγουμε από το 5%. Εδώ πέρα νομίζω πρέπει ακριβώς να δραστηριοποιηθεί ο εισηγητής για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μόρτεν Μέσερσμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές και τον κύριο Τάγκ εισηγητής ο δικός μου γιατί εγώ καλύπτω τις ε, τίτλοποιήσεις. Καλό είναι ότι προχωράμε στις πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Προσπαθούμε ακόμα να τις αναλύσουμε όλες και ιδιαίτερα τις τελευταίες προτάσεις σας. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, όπου απέχουμε. Θέλω κι εγώ, όπως και εσείς, να έχουμε μια ευρύτατη συμμαχία, αλλά επίσης αυτό απαιτεί και κάποια διάθεση συμβιβασμού και βλέπω πως υπάρχουν τουλάχιστον τρία μεγάλα εμπόδια. Η διακράτηση του ρίσκου, όπου δεδομένης της ε, θέλησης ε, και της ε, ικανότητας στο Συμβούλιο να καταλήξουν σε μια καλή και γρήγορη συμφωνία το βρίσκω περίεργο γιατί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς φέρνουμε νέες επίμαχες ιδέες που δεν αντικατοπτρίζουν καμία από τις συζητήσεις μεταξύ των 28 κρατών μελών. Και ούτε η ECB, ούτε η EBA, ούτε η Κομισιόν, ούτε κανένας άλλος δεν ζήτησε κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζονται αυτές οι προτάσεις. Πρέπει απλά να συμφωνήσουμε σε, με, το παγκόσμι, με την παγκόσμια πρωτογραφή. Δεύτερον, για το μηχανισμό υποπτίας. Ίσως ε, να μπορέσουμε να δεχτούμε έναν τέτοιο ρόλο κατευθυντήριο για την ΕΣΜΑ, αλλά η τελική απόφαση βεβαίως επαφίεται στις εθνικές εποπτικές αρχές, δεδομένου του ότι υπάρχουν ακόμα τόσο πολλές διαφορές στη νομοθεσία, τη δομή μεταξύ των κρατών μελών. Και τρίτον, ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα είναι το τι θα γίνει με τα ιστορικά στοιχεία. Ε, σημαντικό για εμάς, ε, σημαντικό για εμάς γιατί είναι σημαντικό για την αγορά. Το σκεπτικό εδώ πέρα δηλαδή είναι να δημιουργήσουμε ασφάλεια για την αγορά και αν δεν βρεθεί ένας ε, τρόπος να αντιμετωπίσουμε ακριβώ αυτά τα παλαιά ιστορικά στοιχεία ενεργητικού δεν θα υπάρξει ασφάλεια. Και δεν θα δημιουργηθεί μετά ανάπτυξη και ε, δουλειέ που είναι ο στόχος αυτής της πρότασης. Οπότε, συμφωνούμε να έχουμε μια ευρύτατη συμφωνία, μια πρόταση με σύνοχη, αλλά πρέπει να ζούμε και στην πραγματικότητα. Οπότε, σας παρακαλώ κύριε Σιγητά, είναι να εγκαταλείψετε όλα αυτά τα όνειρα περί παραδείσου επιγής, να προσγειωθείτε στον πραγματικό κόσμο. Μιλάω για την διακράτηση του ρίσκου, αν δεν έχετε καταλάβει. Και τότε έτσι θα βρεθεί αυτή η πλειοψηφία και θα μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα γρήγορα, με συνέπεια, όπως ακριβώς και το Συμβούλιο. Και νομίζω θα είναι καλό αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Πέτρη Γέζεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επαναλάβω ότι οι αντιρρήσει ε, της Άλντε, οι στόχοι της Άλντε είναι να φτιάξουμε ένα στεναρό πλαίσιο για την απλή ε, τιτλοποίηση στην Ευρώπη, απλή διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πλαίσιο απλής διαφανούς ε, και τυποποιημένης τυφλοποίησης, ούτως ώστε να απομπλοκαριστεί το κεφάλαιο από τις τράπεζες σας και να μπορέσουν να δανείσουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Με αυτά υπόψη υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες ε, για τον κανονισμό αυτό. Θεωρούμε ότι η αντίδραση του εισηγητή με την πρόταση για τη διακράτηση του κινδύνου είναι σημαντική και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα, αλλά μια και το συζήτησαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, ε, περιορίζομαι να πω ότι θεωρούμε ότι η συγκράτηση του κινδύνου θα πρέπει να διατηρηθεί στο 5% ούτω ώστε το STS ε, να είναι βιώσιμο. Ε, με τις άλλες τροπολογίες μας προσπαθούμε να κάνουμε το καθεστώς πιο ευέλικτο και λειτουργικό. Ε, Επομένω, για τις νόμιμες ε, ε, συναλλαγές και τις διατάξεις grandfathering είμαστε πιο ευέλικτοι. Για τις συναλλαγές ABCP η πρόταση της Κομισιόν για τη διάρκεια είναι πολύ περιοριστική και θέλουμε να βάλουμε και τα, και τα και να αυξήσουμε την διάρκεια ε, στα τρία και 6 χρόνια. Για την πιστοποίηση πιστεύω ότι η πιστοποίηση των τρίτων μερών ε, εξασφαλίζει, βάζει και ένα επιπλέον στρώμα ε, ασφάλειας ότι τα κριτήρια του STS πληρούνται. Θέλω λοιπόν να υπάρχει πιστοποίηση των τρίτων μερών με την επιφύλαξη όμως ότι θα πρέπει η μεταβιβάζουσα οντότητα να, έχουν, ε, να έχει πάντα την ε, ευθύνη για την υλοποίηση που έχει εκδοθεί. Τέλος για τη διαφάνεια. Σημερίζομαι τους στόχου του εισηγητή να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε για του επενδυτέ. Όμως θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το μέτρο ε, για να υλοποιήσει αυτό το στόχο είναι αποτελεσματικό. δηλαδή το κόστο του σε σχέση με το όφελό του είναι σωστό. Επίσης να μειώσουμε το βάρος που βάζουμε στις εποπτικές αρχές. Για αυτούς τους λόγους είμαστε προσεκτικοί για την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού αποθετηρίου τίτλοποίησης, όπως προτείνει ε, ο εισηγητής και δεν ξέρουμε αν είναι σωστό αυτό. Ε, περιμένουμε την περαιτέρω συζήτηση και με τους εισηγητές και με τους κοιότητες εισηγητές και ελπίζω να προχωρήσουμε ούτω ώστε να ψηφίσουμε πριν από τις 10 Νοεμβρίου. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ, κύριος Βιέγκας. Ευχαριστώ. Μήνες συζητήσαμε αυτό το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν πιστήκαμε ακόμα για τα πλεονεκτήματα της τυκλοποίησης. Δεν καταλάβουμε ακόμη πώς μέσω αυτής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας θα καταφέρουμε να μετριάσουμε τους κινδύνους των προϊόντων αυτών που ξέρουμε ότι ήταν και στο επίκεντρο της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ξεκολουθούμε να μην θεωρούμε ότι είναι απλά η διαφανή αυτά τα προϊόντα. Δεν έχουμε πιστεί του ναντίον. Ούτε έχουμε πιστεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη ζήτησης. Είναι χαμηλή ζήτηση λόγω των πολιτικών λιτότητας. Όμως, μοχλός της ανάκαμψης δεν μπορεί παρά να είναι η ζήτηση. Εμεί δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια επένδυση στην πραγματική οικονομία, αλλά τι λειτουργίε του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Ε, και αυτό το είδο τα προϊόντα δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι η τιτλοποίηση χρέου είναι ένα είδο ε, να καθαρίσει του ολογισμούς των τραπεζών. Αλλά δεν πρόκειται να φέρει καμιά διαφάνεια στην αγορά. Το αντίθετο. Άρα θεωρούμε ότι ο κόσμος μπορεί, μπορεί πολύ καλά να ζήσει χωρίς τις τηλεοποιήσεις. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα η χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι σημαντικό, πράγματι. Άρα, επειδή είναι σημαντικό το θέμα, δεν θα πρέπει να το αφήσουμε αποκλειστικά στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή είναι η λύση. Δημόσιος έλεγχος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό θα δώσει διαφάνεια αποτελεσματικότητα και χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας. Επομένως, Για τους λόγους που μόλις σας εξήγησα είναι κάπως διαφορετική η θέση μας. Δεν θέλουμε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός, παραπάνω βήματα στη λάθος κατεύθυνση, στην κατεύθυνση που οδήγησε στην κρίση του 7 και 8. Μας ανησυχεί αυτό το νέο κύμα απορρίθμισης και απελευθέρωση. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Μας τα έχει δείξει και η ιστορία. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους τώρα. Ευχαριστώ. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και με τους Σκιώδης ε, έχουμε μια καλή συνεργασία. Μέχρι στιγμής ξέρουμε που διαφωνούμε. Ελπίζω αύριο όταν ξανασταθούμε να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα. Εν είδης να πω ότι αυτό που ανησυχεί κυρίως ε, τους ε, πρασίνωση είναι ότι αυτό το ποιοτικό σήμα αισθιά πρέπει να παραμείνει έτσι, ε, ω τέτοιο. Αν συμφωνούμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα ευρύ ορισμός, αλλά δεν θεωρίζεται ένα ευρύ τμήμα της αγοράς ε, για το οποίο δεν υπάρχει αρμοδιότητα, άρα θα υπομονωμευθούν ε, οι στόχοι της Κομισιόν και οι στόχοι αυτού του προγράμματος. Άλλωστε, θα μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει διπλοποιήσεις, όχι εστίες. Το θέμα είναι εμείς να δούμε Πού δίνουμε αυτή ε, την ε, μάρκα ποιότητα, αυτό το σήμα ποιότητας. Ε, αυτά εισαγωγικά. Τώρα, δύο πτυχέ συγκεκριμένα. Απλούστευση και διακράτηση κινδύνου. Πρώτον, θεωρούμε ότι ο ακριβή ορισμός του ομογενούς, ομοιογενού, θα έπρεπε να γίνει στην νομοθεσία επίπεδο 2 και εδώ θα πρέπει να ορίσουμε τις αρχές όπως είναι συμβατικά, χαρακτηριστικά κτλ. Και δεν θα πρέπει να εστιάζουμε σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο υποκείμενης έκθεση. Επίσης, και άλλα θέματα πρέπει να δούμε. Τράνσινγκ, οι δόσεις, η, ο διαχωρισμός ε, σε μικρότερες δόσεις. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα των τμήματων τιτλοποίησης και πρώτα θα χαθεί η εμπιστοσύνη στα τελικά προϊόντα, στις τελικές αυτές φάσεις. Όμως η βασική απέτηση είναι ε, να εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή η αγορά, τετλοποίηση STS. Επίσης, πρώτη απόπειρα. Πώς μπορούμε να βάλουμε συνθετικά προϊόντα κάτω από αυτή την ε, ταμπέλα. Και πάλι βέβαια μπορούν όποιοι θέλουν να παράξουν συνθετικά παιδιά, αλλά δεν θα έχουν αυτή την, ε, αυτό το σήμα. Δεν θα πρέπει να επεκτείνουμε τον ορισμό. Θα πρέπει πρώτα να γίνει επιτόπια δουλειά από την Κομισιόν. Τώρα, στο δεύτερο θέμα, διακράτηση κινδύνου. Νομίζω ότι η πρόταση βοηθήσει, θα βοηθήσει να γεφυρωθούν οι διαφορές με τις άλλες πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο Seasoning loans, όπως τα λέμε, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. με τις διατάξεις ε, δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Τρεις ε, βελτιώσεις βλέπω εγώ. Μέγιστη διακράτηση, ελάχιστη διακράτηση και βέλτιστο επίπεδο seasoning για να έχουμε το χαμηλότερο συντελεστή δεκάτη κινδύνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες στη συζήτηση που πιστεύουν λίγο πολύ ότι το ίδιο θα πρέπει να είναι το μέγιστο και το ανώ, κατώτερο επίπεδο 5% και 0% το seasoning, το βέλτιστο επίπεδο. Και υπάρχουν άλλες τρεις ομάδες που πιστεύουν ότι μέγιστο ε, και ελάχιστο ποσοστό θα πρέπει να είναι 20-25 και 0 το βέλτιστο. Εμείς προτείνουμε ως πράσινοι το κατώτατο να είναι 10% και 25% το μέγιστο και τα επέδα season 50%. Χαιρόμαστε που βλέπουμε στην τελευταία συμβιβαστική ότι ο συγκεκριτής δέχεται αυτή την προσέγγιση. 20% το μέγιστο και 10% το ελάχιστο και 5% το optimal seasoning. Καλός είναι αυτός ε, ο τρόπος να γεφυρώσουμε τις διαφορές μεταξύ των ε, ομάδων. Και ελπίζω οι σκιώδεις να δουν ε, με ευνοϊκό μάτι αυτή την προσπάθεια συμβιβασμού. Thank you, Marco Valli. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τους δύο εισηγητές για τις προτάσεις αυτές και του Σκιώδη. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Σνάφο Γέγκα για το ότι οι προτάσει αυτές δεν πάνε στην πολιτική κατεύθυνση την οποία θα θέλαμε. Έχουμε να λάβουμε υπόψη να... Τι Τις της αγοράς και πώς όμως θα διαχειριστούμε τελικά τη ζήτηση σε σχέση με τις πολιτικές λιτότητες, οι οποίες κατοχυρώνονται και με τις συνθήκες. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, λοιπόν, μεταξύ της λιτότητας ως αυτό σκοπό και της λιτότητας ε, που σχετίζεται με το ευρώ και δεν έχει συζητηθεί πολύ και προβλέπεται όπως είπα τις συνθήκες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε, να κάνουμε τις προσπάθειες μας να βελτιώσουμε την ε, πρόταση κυρίως θέλοντας να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές. Είπε ε, κάποιος ότι δεν θέλουμε συνθετικά για τελοποίησης STS. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη τυλοποίηση αυτή της Αυτό θα πρέπει να είναι τελευταίο, ε, η έσχατη λύση Επίσης ε, αποκλείσαμε την ε, τηλεοποίηση μέσω τρίτων χωρών. Έχει συζητήσει πάρα πολύ το Κοινοβούλιο για το θέμα της ε, διαφάνειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ειδικά όσον αφορά χώρες offshore. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση για την απλή διαφανή και τυποποιημένη τίτλοποίηση όσον αφορά την σταθερότητα των χρηματαγορών παρατηρώντας και παρακολουθώντας συνολικά και ενοποιημένα δεδομένα. Όσον αφορά τώρα τις εκθέσεις ε, για τις ε, τιτλοποίησεις αυτές, ε, θέλουμε να επιδείξουμε ένα πνεύμα συνεργασίας και θα προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς έχουμε, όπως είπα, ένα πνεύμα συνεργασίας ε, με αυτές τις προτάσεις για να μην καταλήξουμε να πλήξουμε τον κλάδο από τις προτάσεις αυτές. Χρειάζεται όμως αυτή η πρόκληση για να ε, καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα θετικό το οποίο δεν θα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη λύση. Για το θέμα τώρα του συναδέλφου Τζάλμπα ζητήσαμε ακριβώς να υπάρξει μια τυποποιημένη μέθοδος η οποία θα αφορά ε, ακριβώς τις απλές ε, διαφανείς και, τυποποιημένες, ε, και τυποποιημένες τυτλοποιήσεις και πρέπει ακριβώς να διατηρηθεί το όριο θεωρούμε διακράτησης του ρίσκου στο 15% και όσον αφορά τέλος τα συνθετικά αυτά προϊόντα ε, εξορισμού δεν είναι απλά και διάφανα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση και για αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την σχέση μεταξύ αυτών των προϊόντων και της πραγματικής ε, οικονομίας. Οπότε, ελπίζω στην περίπτωση αυτή να επιδείξουμε συνεργασία για να ωφελήσουμε, όπως είπα, και τον κλάδο και τους πολίτες, γιατί το Κοινοβούλιο σε αντίθεση με τα θεσμικά όργανα τα οποία λειτουργούν και κλεισμένων των θυρών θα πρέπει ακριβώ να λαμβάνει υπόψη περισσότερο τα συμφέροντα των πολιτών και του συστημικού κινδύνους. Και να βελτιώσει την κατάσταση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν βλέπω τον κύριο Μινιός. Περνάμε λοιπόν στον σκιώδη εισηγητή, τον ε, κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς κύριε Σιγητά, κύριε Θάλβα και με βέβαια και τους άλλους ε, σκιώδη ε, Σε πολλές ε, συναντήσεις που είχαμε προσπαθήσαμε να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με τις αρχικές μας θέσεις και κάποιοι εξημών να εξακολουθούμε να εμένουμε σε αυτές τις θέσεις. Θέλουμε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο αυτή η διαπραγμάτευση που δεν το βλέπουμε να συμβαίνει μέχρι τώρα. Ποια είναι τα πιο επίμαχα για τις κεφαλακές απαιτήσει. Τέσσερα σημεία. Πρώτον, η σχέση των απαιτήσεων για τις ε, τιτλοποίησεις αιστείες αυτές που θα μπορούσαν να τύχουν αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης στο τέφα της τις απαιτήσεις. Και εγώ νομίζω ότι η πρόταση ως έχει αυτή η συμβαστική πρόταση που συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρία των συντονιστών ουσιαστικά υποβαθμίζει σημαντικά τις απαιτήσει αρχικής πρότασης κομισιών Και η δική μου πολιτική ομάδα στο συγκεκριμένο εδάφιο πράγματι δεν είχε καταθέσει ε, και μια σειρά τροπολογιών, σημαντικών τροπολογιών, γιατί ουσιαστικά συμφωνούσαμε με την πρόταση της Κομισιόν. Επομένως, ε, ο συμβιβασμό στο βαθμό που, όπως είπα, υποβαθμίζει και κατά την άποψή μου σημαντικά τις απαιτήσει ε, που επιβάλλονται στις τυπλοποιήσεις τις απλές διαφανείς και τυποποιημένες, ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είναι αρκετά μακριά από τις δικές μας θέσεις αυτός ο συμβιβασμός. Πέραν αυτού, θέλουμε να συζητηθεί το θέμα της ιεράρχησης ε, για τις κεφαλαίκες απαιτήσει. Για το θέμα αυτό έχουμε καταθέσει τροπολογίες, ούτω ώστε η και αξιολόγησης να μην μολύνουν, αν θέλετε, την νομοθετική διαδικασία κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν οίκους αξιολόγησης και αξιολογήσεις να μείνουν εκτός του συστήματος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τουλάχιστον για τις ε, STS, ε, αλλά και για το σύνολο των τυπλοποιήσεων ή δυνατών. Αυτή είναι η άποψή μας και θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε την επίσημη ε, τοποθέτηση του εισηγητή, ελπίζοντας, όπως είπα, αυτοί και οι αξιολές να μείνουν εκτός της νομοθετικής διαδικασίας. Και έτσι πιστεύω θα βελτιώσουμε ε, την ολοκλήρωση και συνοχή της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση της Κομισιόν τώρα εισάγει σε ένα άρθρο στο τέλος του κειμένου και με ένα περιορισμένο τρόπο το ότι οι συνθετικές θυλοποίησεις θα μπορούσαν να έχουν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση και απαιτήσει. Η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε πολύ πιο προσεκτικά αυτέ τι συνθετικέ τυπλοποιήσει, ποιες θα, τι θα μπορούσαν να είναι ακριβώ. Και εμεί πιστεύουμε ότι η Κομισιόν πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία και να καταθέσει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκρινίζει και θα διασκεδάσει τι ασάφει και τι αβεβαιότητε για τι συνθετικέ οι που θα μπορούσαν να πάρουν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση. Να είναι δηλαδή λιγότερε κεφαλικέ απαιτήσει. Γιατί φαίνεται ότι δημιουργούμε αυτέ τι αιστείε, δημιουργούμε τι τιτλοποιήσει με λιγότερε κεφαλικέ απαιτήσει και έπειτα στο τέλο έχουμε ε, μια διαφορετική ομάδα τιτλοποιήσεων που δεν θα πρέπει να τηρήσουν παρά κάποιε από τι κεφαλικέ απαιτήσει και όχι άλλε ε, κτλ. κτλ. Τέλος η ομάδα μου κατέθεσε τροπολογίες για την αναθεώρηση των ε, κεφαλαίων απαιτήσεων, τον πυρήνα δηλαδή, διότι θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση έχει απόλυτη σχέση με την έκθεση του Πολ Τάνκ που δημιουργεί αυτές τις τετλοποιήσεις STS. Άρα στο βαθμό που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ε, πραγματικά ε, απλές διαφανή και τυποποιημένη τυλοποίηση, ναι, θα μπορούσαμε να δεχθούμε την πρόταση Κομισιόν για τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει. Αλλά αν αυτέ οι αιστείε δεν είναι όσο διαφανεί θα θέλαμε, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να δούμε και λίγο καλύτερα τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών αγώνων. Αυτού του δύο κανονισμού, λοιπόν, όπω και με οποιονδήποτε άλλο ε, χρηματοπιστωτικό κανονισμό, ε, θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, ασφάλεια Είπε και ο Τμαρκάρας ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο που θα πρέπει να είναι ταχύ, αλλά θα πρέπει να είναι και ασφαλές. Άρα θα πρέπει να, να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την ασφάλεια με την ταχύτητα. Μείωση κινδύνου για την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, Πάμπλο. Κοιτάξτε, εμεί ε, σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε με τον εισηγητή εδώ πέρα και ελπίζουμε να διατηρηθεί η κατεύθυνση την οποία έχει. Όμως κάτι το οποίο θίξαμε και ε, θίξε και οι Άλτε στην τροπολογία 159 αφορά ακριβώς το θέμα της λήξης. Δεν θεωρούμε ότι είναι αυτό το σωστό μοντέλο για τον υπολογισμό. Επίσης, το ότι δεν υπάρχει διαφθορά μεταξύ των ε, δόσεων ε, εκείνων οι οποίες είναι, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ε, άλλες. Επίσης, το ECR έχει υποβάλει μια τροπολογία την 174 για ξεκάθαρες ε, προδιαγραφές ε, των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τον ε, υπολογισμό και την χρήση των κατάλληλων δεδομένων. Υποστηρίζουμε ακριβώς τις ίσες ευκαιρίες αλλά και την ίση εποπτεία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές συνεχώς. Όσον αφορά τέλος την ιεραρχία των μεθόδων, υπήρξαν κάποιες τροπολογίες που κατατέθηκαν. Γνωρίζω επίσης ε, τα όσα είπε ο εισηγητής για τις εξωτερικές ε, αξιολογήσεις. Όμως ε, βεβαίως συμφωνούμε και με άλλες απόψεις της Άλντε όσον αφορά ακριβώς τα εμπορικά αυτά χρεόγραφα με τα καλυμμένα με στοιχεία ενεργητικού. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε μια συνένεση για να υπάρξει, να υπάρξουν κάποιοι νόροι στην χρήση των ERBA. Τέλος, ε, δεν συμφωνούμε με όλες τις ε, αναθεωρήσεις. Θέλουμε μόνο την τυποποιημένη μέθοδο. Επιπλέον, αν μου επιτρέπετε να γίνω κάπως πιο συγκεκριμένο, το ECR δεν υποστηρίζει τροπολογίες 122 και 123 στο άρθρο 250 που αφορά μια άρρητη στήριξη. Θεωρούμε βεβαίως ότι θα πρέπει ακριβώς να αποτελεί τμήμα της αξιολόγησης, αλλά έτσι υπονοούμε ότι αυτά τα προϊόντα εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Και βεβαίως τίθεται το ζήτημα του τι ακριβώς σημαίνει στήριξη. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πως μια συναλλαγή η οποία έχει γίνει με μια δίκαιη τιμή στην αγορά δεν ε, υφίσταται ακριβώς ε, αυτή την στήριξη και θα ήθελα να συναντήσω και τους υπόλοιπους σκιοδησηγητές και να μένω τη συζήτηση μαζί τους. Και τους ευχαριστώ για την επικοδομητική ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ, Μάικλ Τόιρερ. Äh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σάλμπα και τον κύριο συνδέονται τα δύο θέματα. Έχω την εντύπωση πως ε, έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο. για να μπορέσει να δοθεί μια νέα όθηση στην πραγματική οικονομία χωρίς βεβαίω να αναλάβουμε ξανά τους κινδύνους οι οποίοι υπήρχαν στο παρελθόν. Έχουμε ακριβώς τις προτάσεις συμβαστικών ε, τροπολογιών που κυκλοφορούν. Θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Αν δούμε την σημασία για την πραγματική οικονομία, έχουμε ακριβώς τα asset-backed commercial papers, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στη leasing αυτοκινήτων, αλλά και σε άλλα μοντέλα χρηματοδότησης πραγματικής οικονομίας. Και εδώ πέρα προέκυψε ότι σε σχέση με την πρόταση της ε, Κομισιόν και τις άλλες ε, διατυπώσεις, υπάρχει το πρόβλημα ότι αν ε, δεν υπάρχει ο διαχειριστής, ταυτόχρονα δεν υπάρχει πια και η μέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης, κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να το δεχτούμε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε υποβάλει μια πρόταση για το πώς ε, θα μπορούσαν ε, να διατηρηθούν και στο μέλλον οι προσεγγίσεις αυτές εσωτερικής αξιολόγησης, γιατί έχω την εντύπωση στις ε, συζητήσεις πως όλες οι πολιτικές ομάδες ε, δεν θέλει να, καμία ομάδα δεν θέλει να δυσκολέψει αυτά τα asset back commercial papers. Αντιθέτως θέλουμε οι τίτλοποιήσεις ε, να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Από το βασικό σημείο πρέπει να είναι να ξεκινήσει ξανά η αγορά των τίτλοποιήσεων χωρίς να υπάρξουν ακριβώς όλα αυτά τα φαινόμενα που είχαν τις αρνητικές επιπτώσεις στο παρελθόν. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Viegas. Όχι. τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ε, είμαι στην ε, προνομιούχα θέση να είμαι ε, συγκίτρια και για τα δύο θέματα. Τυχερή που είμαι. Εισαγωγικά, η θέση μας είναι ότι η καρδιά του, του σχεδιασμού του STS θα πρέπει να είναι ε, ένας νόμος που θα καλύπτει και, την, και το άλλο θέμα που συζητάμε στην Επιτροπή. Γιατί αυτό που συζητάμε τώρα είναι δευτερεύον θέμα. Επίσης, η μείωση των, απαιτήσεων, ε, των προληπτικών απαιτήσεων ε, θα πρέπει να μας δώσει μία τελείως διαφορετική αγορά. Ε, καταρχάς, όταν μία τράπεζα επενδύει στην διδοποίηση μιας άλλης τράπεζας, θα πρέπει να ε, εφαρμόζει ψηλότερη στάθμιση ε, για να δει εάν υπάρχει συστημικός κίνδυνος και για να υπάρχει ε, διασπρά του κινδύνου σε όλους τους τομείς. Δεύτερον, δεν έχει νόημα να, γίνει, να δώσουμε ειδική εξαίρεση για τη σύνθετη τυπλοποίηση, ακόμα και στα πλαίσια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ορισμένε περιπτώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιε μικρομεσαίε επιχειρήσει εμποδίζονται ε, πολύ λόγω τη έλλειψη πίστοση, αλλά δεν είναι αυτό γενικό πρόβλημα. θα ήταν λάθο να χαλαρώσουμε του κανόνε τη τυπλοποίηση και να ε, σπάσουμε αυτή τη διάξη που υπάρχει ανάμεσα στην ε, τυπλοποίηση STS και μη STS. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αναζητήσουν να, τη λύση του προβλήματό τους στην, στην Έχουμε ε, Επίσης, τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις από τράπεζες για την ίδια συναλλαγή. Οι νομοθέτες μπορούν να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ε, και να είναι απλή ε, και τυποποιημένη η τιτλοποίηση. Εάν ε, πρόκειται για STS, όντως πραγματική STS, τότε θα πρέπει να έχουμε μια κλασική τιτλοποίηση, πραγματική κλασική τιτλοποίηση. Εγώ έχω παρέμβει, λέει ο κ. Επομένως δεν χρειάζεται να ξαναπάρω τον λόγο. Από το ΙΕΝΕΦ, ουδής, οι συγκητές μας, πρώτα απ' όλα ο κύριο Τάγκ. Έχω ένα ομιλητή για το ΚΑΤΣΙΑΙ. Έχουμε χρόνο. Πολύ σύντομα. Η ανησυχία μου αφορά το, την αντίληψη που έχει το Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Ξέρω πόσο περίπλοκα είναι. Ε, γίνονται τεράστιες συζητήσεις, πολλές τροπολογίες, αλλά θα πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος έξω από εδώ περιμένει το Κοινοβούλιο να κάνει κάτι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η τηλεοποίηση είναι τμήμα ενός μεγάλου εγχειρήματος μιας μεγάλης ε, ένωσης κεφαλαιογορών. Όταν ανακοινώνετε με την πανοκρουσία, ότι θα φτιάξετε μία ένωση αγορών και τελικά έχετε μόνο τιτλοποίηση και για κάποια θέματα διέξοδο, μην ξεχνάτε ότι άλλοι στο απ' έξω μας παρατηρούν. Και δεν θα πρέπει να γίνουμε όμοιροι των εξελίξεων στο Ενωμένο Βασίλειο και των δικών μας εσωτερικών ιδεολογικών διαφορών, γιατί τελικά θα χάσουμε όλοι μας. Ευχαριστώ. Άλλοι ομιλητές. Όχι. Ο κ. Στάγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για το τελευταίο σημείο. Όντω είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι, όχι μόνο για αυτό το φάκελο, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η Τραπεζική Ένωση. Και αυτό το θέμα είναι αμφίμαχο, επίμαχο μάλλον, αλλά χρειάζεται και εκεί να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε, να δώσουμε κάτι το χειροπιαστό. θα πρέπει αυτό, για να πετύχουμε αυτό που λέτε, να είναι διατεθειμένες οι πολιτικές ομάδες να συμβιβαστούν. Αυτό που έδειξε αυτή η ανταλλαγή απόψεων δείχνει ότι υπάρχει επικοδομητικό πνεύμα. Και ο Παύλο Θάλμπα ε, έχει επικοδομητική στάση, τον ευχαριστώ και οι υπόλοιποι σκιώδεις ε, το ίδιο και αυτό είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε αποτελέσματα. Ε, όμως υπάρχουν κάποια θέματα που τα έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και περιμένω. Ε, όχι αυτό που είπες Μόρτεν, ε, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε σαν πρόβατα το Συμβούλιο. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία για να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για την τυλοποίηση. Γιατί αλλιώς θα είμαστε μια τεχνική ένωση η οποία δεν θα τη χάνει υποστήριξη από κανέναν. Δεν έχει νόημα να έχουμε μια μικρή πλειοψηφία. Θέλουμε αυτά τα προϊόντα να είναι καλύτερα από, τα, από, αυτά που ήταν, από αυτά που είχαμε στο παρελθόν για να δείξουμε στον κόσμο ότι πραγματικά μάθαμε το μάθημά μας. Αυτό θέλω να πετύχουμε, θα χρειαστεί χρόνος. Ε, θέλω επικοδομητική προσέγγιση, γι' αυτό χρειαζόμαστε και συνεπείς προτάσεις. Οτιδήποτε προκύψει από εμά θα πρέπει να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό. Θα πρέπει να δουλεύει. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και με, συμφωνώ με τον Όκμαρ ότι είναι σημαντικό θέμα, είναι το θέμα της ε, συγκράτησης του κινδύνου. είναι, ποια είναι η απάντηση, 5, 25%, όχι, 15% λέμε. Ε, αν θέλετε, λέω στις πολιτικές ομάδες, να κάνετε κάτι, ε, να έχετε καλές ιδέες, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις δύο πλευρές, και τις ανησυχίες και των δύο πλευρών. Μέχρι στιγμή ήμασταν επικοδομητικοί. Πρέπει να συνεχίσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Το χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πλατή, ε, σε ένα συμβιβασμό μάλλον με πλατιά συνένεση. Ο κύριος Θάλμπα. Ο Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, ακόμη αρκετά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Πάντω κάνουμε καλή δουλειά γιατί προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ προτάσεις. Υπάρχουν και κάποιες κοινέ ανησυχίε για τη σύνδετη τυλοποίηση παραδείγματι. Όλοι συμφωνούμε πιστεύω πως ε, και εμείς πρέπει να διδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά με τη σύνθετη στην θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση, ναι, πράγματι όλοι ανησυχούμε για τον ρόλο των οίκων αξιολόγησης και νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο υπάρχει δική μου πρόταση, υπάρχει η άλλη πρόταση και πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Τέλος, <clears throat> συμφωνώ πως ανησυχεί η κοινή γνώμη για το τι κάνουμε. Ξέρετε όμως, το θέμα είναι άκρος τεχνικό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχυση στην κοινή γνώμη. Το αντίθετο πρέπει να καθησυχάσουμε την κοινή γνώμη, να τους δώσουμε, αν θέλετε, μια βεβαιότητα, μια σιγουριά. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χαθεί αυτό το στίγμα που φέρουν πάνω τους αυτές τις κλοποιήσεις, ότι οφείλονται σε αυτές τις κρίσεις και τα λοιπά. Πρέπει να τους πείσουμε ότι χρειάζεται τυπλοποίηση για να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ που όπως είπα ακριβώς είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. δεν μπορούμε βέβαια να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το καταλάβουν 100% από μόνοι τους ε, οι συμπολίτες μας. Πρέπει να τους δώσουμε λύσεις, πρέπει να τους βοηθήσουμε ε, να καταλάβουν αυτές τις πολυτεχνικές εκθέσεις. Και ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις ε, ώστε η κοινή γνώμη να τα καταλάβει όλα αυτά που λέμε και να μην προκληθεί σύγχυση στον κόσμο για το τι κάνουμε εμείς εδώ. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Θέλω να υπογραμμίσω ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν θέματα, ιδίως ένα, βλέπω να δημιουργεί πολλές διαφωνίες, δεν υποτιμώ τη σημασία των διαφόρων θεμάτων και τις διαφορές, αλλά νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμες οι αποκλήσεις απόψεων και ο έχετε κάνει ήδη πολλά για να εντοπίσει οι κοινέ λύσεις, άρα προχωρούμε, δουλεύουμε. Μας μένει ένας μήνας πριν την ψηφοφορία. Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτός ο μήνας ε, θα αξιοποιηθεί τα μάλα για να γίνουν συζητήσεις, να βρεθούν λύσεις και πράγματι να καταφέρουμε να στηρίξει αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία για να ολοκληρωθεί η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή και έτσι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον τεμέρι διάλογο. Άρα είναι ώρα για δουλειά πολύ νωρί. Για να πούμε ότι πετύχαμε ή ότι τα έχουμε καταφέρει, σε καμία περίπτωση δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Καλή δουλειά λοιπόν στην Ευρωκοινευτική Ομάδα και είμαι βέβαιος ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα προσπαθήσουν να συνεισφέρουν και να δώσουν την υποστήριξή τους ε, και τις προτάσεις. Γιατί γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το ε, θέμα, αυτή η νομοθετική πρόταση. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο εξέταση των τροπολογιών της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής, εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016. Άλφρεντ Σαντ είναι συγητής. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, Θέλω να ευχαριστήσω τους και ηγητές, ε, τους βοηθούς, το προσωπικό που συνεργάζονται, ε, που συνεργάστηκαν ώστε να έχουμε αυτή την έκθεση. Βέβαια, ε, αν ε, υπάρχουν ελαττώματα σε αυτήν την έκθεση, έχω την πλήρη ευθύνη εγώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το έτος σε σχέση με τις προτάσεις της τάσης αναχώρησης της Κομισιόν, έχω να κάνω κάποιες προτάσεις και καταλήγω σε κάποια συμπεράσματα και το λέω πείτε σε κάποιοι. Μείωση τη συστάση τη Κομισιόν, καλύτερο αυτό για να έχουν καλύτερο αντίκτυπο, γιατί αλλιώ υπάρχει σύγχυση και παραγνωρίζονται κάποιε. Για την εκπόνηση τη έκθεση μου με τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε και τι λοιπέ τροπολογίε, στόχο είναι ο εξορθολογισμό τη παρουσίαση και εστιάζουμε σε επενδύσει, σε ένα θέμα μόνο. 330 τροπολογίε Θέλουμε να βρούμε ένα κοινό κείμενο. Ο στόχος μετριάζεται λοιπόν. Ελπίζω να μην έχει αλλοιωθεί πολύ. Μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Πάντως νομίζω ότι ε, τα βασικά επίπεδα, τα βασικά ζητήματα παραμένουν. Άλλες εξελίξεις ε, από για τις περιφέρειες, νότος ε, κτλ. έχουμε το δίλημα των οικονομιών της Ευρωζώνης ε, περισσότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είναι ένα κεντρικό δίλημα για τις καπιταλιστικές οικονομίες. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ συνεδρίασε με το διοικητή της Γαλλικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Γαλλίας, τον κύριο Ντεγκουαγιό, που στην παρουσίασή του τόνισε το επενδυτικό έλλειμμα που μαστίζει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, παρά το χαμηλό κεφαλαίου και είπε ότι ο λόγος είναι δυσνόητος. Γι' αυτό και δεν έχουμε μεγάλα ποσοστά ανάπτυξη. Όλοι πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα και να εστιάσουμε στο πώ μπορούμε αυτή την απροθυμία για επενδύσει να την αναστρέψουμε. Υπήρξε ένα επιχείρημα που ακούς και συζητήσει ότι το μόνο επιτόκιο που κάλυπτε και πολλές ε, διαφορετικές καταστάσεις, ε, ίσως να είναι ένα πρόβλημα το ενιαίο πτώκιο. Πρέπει να αναζωογονήσουμε την επενδυτική όρεξη. Αλλά με το τρέχον σύστημα στην Ευρωζώνη δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Όμως δεν εξηγεί γιατί και στην Αμερική η οικονομία έχουμε αυτά τα τόσο ιστορικά χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και στην Ευρωζώνη. Κατά το παρελθόν υπήρχαν περίοδοι που ήταν πολύ ψηλότερα τα σημερινά τα επίπεδα επενδάσεων επενδύσεων. Παρότι δεν λειτουργούσε στο βάλιστο επίπεδο ευρωζών. Πιστεύουμε ότι είναι καλό και σκόπιμο να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τα παλιά καλά επίπεδα επενδύσεων. Και όλες οι ομάδες θα πρέπει να συμφωνήσουν για τις επενδύσεις. Ε, είτε είναι δυτικές, είτε δημόσιες και είτε κάτι άλλο. Ε, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία εύση ε, Τη στηρίζουμε όλοι, απλά δεν εκτιμούμε με τον ίδιο τρόπο το πόσο αποτελεσματική. Πάντως στηρίζουμε τη διεύρυνσή της και επέκτασή της αυτής της πρωτοβουλίας, αυτού του ταμείου. Σε ό,τι αφορά τις ε, ειδικέ συστάσεις αναχώρα, βλέπουμε χαμηλές, χαμηλά ποσοστά εφαρμογής αυτών των συστάσεων. Θα πρέπει να δούμε περισσότερο λοιπόν αυτά τα θέματα. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ τη ευρωκεντρική προσέγγισης τη Κομισιόν και των εθνικών προοπτικών. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, άρα εδώ θα έχουμε μία αντιπαραβολή απόψεων και καλό είναι να θυσιάσουμε κάπου τα εθνικά συμφέροντα για πανευρωπαϊκές στρατηγικές. Να δώσουμε κάποια εργαλεία υπάρχουν κάποιες τάσεις ε, φυγόκεντρες και αυτές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν και υπο... οι αρχές περιφερειακές, ε, οι υποεθνικές, που και αυτές ευθύνονται κατά κάποιο τρόπο για το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων. Στο σχέδιο έκθεσης αυτές οι αρχές ε, αναγνωρίζονται ότι έχουν ρόλο και για την υλοποίηση των συστάσεων αναχωρών. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν περισσότερο ρόλο για να υπάρχει μεγαλύτερη διοκτησία και λιγότερο ε, χάσμα σε σχέση με τις Βρυξέλλες και στο τι υιοθετείται σε εθνικό επίπεδο για να εκπληρωθούν και απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, και βεβαίως ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική πολιτική της Ένωσης διαφέρει από ομάδα σε ομάδα. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε το οικονομικό μοντέλο, αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε το πιο επιτυχημένο, την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Πρέπει επίσης να προσέξουμε οι συστάσεις αναχώρα να μην αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης, ε, δηλαδή πράγματα τα οποία μας αρέσουν να μην ε, ασκούμε καμία κριτική και το αντιστροφό οι συστάσεις αναχώρα έχουν ε, ως αποστολή ακριβώς να προσπαθήσουν να αντιστρέψουν λαθασμένες εξελίξεις. Αυτό βεβαίως πετυχαίνει μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα και η διάθεσμες χώρες της να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Γι' αυτό εμείς είχαμε αντίρρηση όσον αφορά το να προσθεθούν στην γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου επιπρόσθετη δείκτες, επιπρόσθετα θέματα τα οποία δεν έχουν ούτε μία σχέση με το αντικείμενο γιατί για εμάς ήταν σημαντικό να δούμε το ποιε είναι οι δομέ οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα προωθούν τις επενδύσεις και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι φιλικό προς τις μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις. και βεβαίως να πάμε προς την κατεύθυνση την οποία προτείνει η ΕΦΣΑ και υπάρχει το μεγάλο ζήτημα των δημοσίων προϋπολογισμών στα κράτη-μέλη. Ένα θέμα το οποίο είναι, εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή των όσων συμφωνούμε μεταξύ μας. Έχουμε πάνω από 160 παραβιάσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ακόμα δεν έχουν υπάρξει σαφείς κυρώσεις ή κάποια μέτρα. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει νομίζω να εργαζόμαστε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων του ακολούθησε αυτόν τον δρόμο. Βεβαίω υπάρχει και κάποια, κάποιος πολιτικός ανταγωνισμός. Και βεβαίως η σύγκληση δεν θα πρέπει να είναι ένα μέσο εξίσωσης ε, και μάλιστα εξίσωσης ε, προς τα κάτω θα πρέπει το μέτρο να είναι η καλύτερη και εκεί να προσανατολίζονται και οι άλλοι. Και κάθε χώρα βεβαίως να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά της ε, πλέον εκτήματα. Βεβαίως χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για τις συμβαστικές τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί έτσι ακριβώς φαίνονται και οι προτεραιότητές μας. Και ελπίζω έτσι τελικά να έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γιώργη Σταρμπάτη. Έχω βεβαίω εξηγήσει ήδη ποιες είναι οι βασικές μας οι αντιρρήσεις. Θα τις υπενθυμίσω. Τα είπε και ο κύριος Φέρμπερ. 160 παραβιάσεις του Συμφώνου Σταθερότητας. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά προβλήματα, θα έλεγα μια διαφωνία, την οποία προσπαθούμε να γεφυρώσουμε μέσω κάποιων συμβιβασμών και μετά διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι δεν τηρούνται οι συμβιβασμοί γιατί οι χώρες ακολουθεί κάθε το συμφέρον της και έτσι θα συνεχίσει να έχουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, η νομισματική ένωση έχει νόημα αν όλες οι χώρες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλιώ διαλύεται. Και βλέπουμε και στο παρελθόν ότι είχαμε νομισματικές ε, ενώσει που διαλύθηκαν και τώρα προσπαθούμε, βλέπουμε ότι οι χώρες ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις και προσπαθούμε να τις συμβιβάσουμε. Ενώ αποδεικνύεται ότι το ευρώ για κάποιες χώρες είναι υποτιμημένο και για άλλες είναι υπερτιμημένο. Και εδώ πέρα συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος λέει από μόνος του ότι δεν είναι ιδανικός χώρος νομισματικής ένωσης η Ευρωζώνη. Ε, βεβαίως η διαφωνία μας είναι ότι ο εισηγητής θεωρεί ότι με κάποια μέτρα οικονομικού συντονισμού ε, θα καταφέρει να ε, ακολουθήσουν οι χώρες μια κοινή πορεία. Ενώ η ομάδα του ECR θεωρεί ότι οι εξελίξεις δείχνουν ότι δεν είναι επιτυχής μια τέτοια πορεία. Και η συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι ότι όταν δεν είναι ενιαία αυτή η πορεία, οι μεν λένε στους δε πρέπει να ακολουθήσετε τη δικιά μας πορεία. Ότι πρέπει ξέρω εγώ να ακολουθήσετε πολιτική λιτότητας, όπως λέει η κυρία Μέρκελ. Όταν χωρίζουν οι δρόμοι, πρέπει ο ένας να προσαρμοστεί στον άλλον από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως οι χώρες δεν το θέλουν αυτό. Και αυτό το δίλημα εμφανίζεται ξανά και ξανά στην νομισματική ένωση. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρη η απέτηση. Θα πρέπει οι χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια πορεία σταθερότητας να έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την Ένωση. Ο καθένας αυτό θα πρότεινε αν δεν υπήρχε το ευρώ. Αλλά επειδή υπάρχει το ευρώ επιμένουμε στο δόγμα ότι πρέπει να το διατηρήσουμε και να κατευθύνουμε την πολιτική μας προς τα Είναι λάθος ο δρόμος, γι' αυτό η ομάδα του ECR προτείνει να υπάρξει ένα δικαίωμα προσωρινής αποχώρησης για τις χώρες για να αποκαταστήσουν την διεθνή τους ανταγωνιστικότητα. Και θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης ταυτόχρονα και ένα κούρεμα κρέους, ε, όπως πρότεινε και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ για την Ελλάδα. Να τους δοθεί δηλαδή μια μεταβατική βοήθεια για να έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Λοιπόν η διαφορά του ECR είναι ότι εμείς δεν επιμένουμε στο δόγμα το οποίο έχει αποδειχθεί λανθασμένο. Πρέπει να δώσουμε την ελευθερία στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να έχουν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο που θα κρατήσει τους νέους στη χώρα και θα μειώσει την ανεργία. Γι' αυτό θέμε και το λέμε, συζητάμε ξανά μήπως θα είναι καλύτερα να δούμε την αλήθεια κατάματα και να πούμε Ε, μήπως για κάποιες χώρες θα ήταν καλύτερο να αποχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τους φιλελεύθερους. Κύριο Στόιερ. Εγώ δεν είμαι σκιώδης εισηγητής, αλλά πω για τους ε, φιλελεύθερους πως η δημιουργία της Ευρωζώνης έχει πλέον εκτήματα μια ενιαία εσωτερική αγορά η οποία βεβαίω έγινε πιο ενοποιημένη με το ευρώ. Στη σταθερότητα βεβαίω υπήρξε μια υποχώρηση την οποία παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία. Ε, δηλαδή υπήρχε μια ολοκλήρωση της αλυσίδας παραγωγής ε, αξίας η οποία όμως υποχώρησε με την οικονομική κρίση. Και το ερώτημα είναι πώς θα έχουμε σε μια νομισματική ένωση μια κοινή οικονομική πολιτική. Γιατί ήταν σαφές ότι θα έπρεπε να υπάρξει και μια πολιτική ένωση μετά την νομισματική ένωση. Και εδώ πέρα έχει κάποιο δίκαιο ο καθηγητής ε, Σταρμπάτη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει μια ενιαία άποψη στα κράτη-μέλη για το τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτή η κοινή οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο πρόβλημα το οποίο αφορά τα πλεονάσματα, τα ε, ελλείμματα και έχουμε την ιδέα ότι μπορούμε μέσω κρατικών παρεμβάσεων και κατευθυνόμενης οικονομίας ε, να μειώσουμε τα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου. χωρίς δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει μέσω της οικονομίας της αγοράς, αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς οι φιλελεύθεροι. Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι πράγματι η ανταγωνιστικότητα, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής. Κάτι το οποίο εμείς δεν βλέπουμε στην τωρινή συζήτηση είναι το πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα, το κενό τεχνολογίας και καινοτομίας. Χωρίς ε, μια υποτίμηση των μισθών που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις χώρες ε, της περιφέρειας. Και επηρεάζει αρνητικά το, τους ε, λαούς. Πώς θα οδηγηθούμε λοιπόν σε ένα περιβάλλον που θα κάνει τις χώρες αυτές ξανά ανταγωνιστικές και ο τομέας αυτός είναι νομίζω υποτιμημένος της συζητήσεις στα κράτη-μέλη. Εν ολίγης, λοιπόν θεωρούμε πως θα πρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας να α, αναζωογονηθεί. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα πως είναι κάτι το οποίο όλοι τηρούν εθελοντικά και θα πρέπει ακριβώς να το τονίσουμε αυτό και θα το τονίσουμε στις απολογίες μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βιέγκας, θέλει το λόγο για την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εγώ θα διαβάσω τις σημειώσεις της συναδέλφου Παλώμα, ε, της συναδέλφου κυρίας Παλώμα, η οποία είναι σε αντιπροσωπεία της Γκουε που έχει επισκεφθεί την Κίνα. Τρεις-τέσσερις ιδέες έχει. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, λέει η κυρία Παλώμα, δεν μπορούν να επιλύσουν την κρίση. Έχουμε ψηλή ανεργία, έχουμε μεγάλη φτώχεια που εξαπλώνεται. Έχουμε τους εργαζόμενους φτωχούς, τους νεόπτωχούς, οι οποίοι πλήττονται λόγω κρίσης, ε, λόγω της μείωσης των ε, μισθών. Και όλα αυτά είναι προϊόν της υποκρισίας. Μοιάζει κάποιες χώρες να αντιμετωπίζουν τη λιτότητα από τη μία, που δεν, τις, ε, δεν τους επιτρέπει να επενδύσουν, και από περικοπές των διαφορετικών ταμείων. Επίσης, οι προτινόμενες ε, περικοπές των διαρθρωτικών ταμείων για την Ισπανία και την Πορτογαλία, από τη μία και οι στόχοι του ευρώ από την άλλη, δεν μπορούν να συγχωνευτούν, δεν μπορούν να παντρευτούν μεταξύ τους. Έχουμε παράλληλα ιδιωτικοποίησεις, καταράκωση του κράτους πρόνοια, τη μεταφορά του βάρους ε, στους εργαζόμενους ε, πιο επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα δηλαδή που περνάει. Αυτό βρίσκεται πίσω από το ευρώ και όλα από όλους τους κανόνες που επιβάλλονται στις διάφορες χώρες. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι την δυνατότητα εκδημοκρατισμού της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω της απόπειρας Εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Αυτή την ιδέα της, ε, του ownership. Ο μόνος τρόπος για να εκδημοκρατικοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια να αποφασίσουν τις πολιτικές τους. Να αποφασίσουν την ανάπτυξη που θέλουν. Αυτά μου είπε η συνάδελφος κυρία Παλώμα. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Η, λέει ο κ. Ούρτασον. Ε, παιδί, έκθεση, ε, εστιάζει η έκθεση στις επενδύσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτό, είναι σωστό. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις ε, στην έρευνα, ε, εκπαίδευση, ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτομία, σωστό αυτό. Τα λέμε αυτά εδώ και χρόνια ότι το μείγμα πολιτική ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να υποστηρίξει τι επενδύσει. Η έκθεση τα λέει αυτά. Δεύτερον, να αποφύγουμε ε, μία κούρσα προ τα κάτω για τα πρότυπα εργασία και του μισθού, σωστό, και όλε οι αναφορέ που κάνει για να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις αυξανόμενε ανισότητε την καταπολέμηση τη φτώχεια. Αυτέ οι αναφορέ είναι πολύ σημαντικέ και υπάρχουν στην έκθεση. Φυσικά θα θέλαμε η έκθεση να αναγνωρίσει την αποτυχία και τα ελλείμματα του τρέχοντος πλαισίου διακυβέρνησης. Καταλαβαίνω όμω τα πλαίσια μια τελική ε, συμφωνία αυτά ήταν δύσκολο να περάσουν στην έκθεση. Αλλά εμεί επιμένουμε. Δύσκολο είναι να βρούμε ένα καλύτερο και πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικής αν κρατήσουμε τα στοιχεία διακυβέρνησης όπως είναι τώρα. Επίσης, δύο, πολλά, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για μας είναι οι συμβιβασμοί D και E. Ε, το ένα αφορά την ανάγκη να κρατήσουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους ε, στις ειδικέ εκτάσεις αναχώρα και η μετάβαση από την ε, φορολόγηση εργασίας στη φορολόγηση του περιβάλλοντος. Μπήκε και αυτό στο συμβασμό. Τώρα όμως έχουμε χωριστές ψηφοφορίες Ελπίζω να μην καταπέσουν αυτά τα δύο στοιχεία και θα ήταν, ε, γιατί είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα μου. Επίσης ε, υπήρχαν στο ψήφισμα πριν από έξι μήνες. Ε, θα υπάρχει πρόβλημα για μας αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην έκθεση. Ευχαριστώ, Μαρκο Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για την δέσμευση και το ζήλο που έχει δείξει για να προσπαθήσει να χτίσει πλατιά συνένεση στο Κοινοβούλιο για αυτή την έκθεση, που είναι πολύ σημαντική. Ε, το πλαίσιο της διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για το Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο ε, και γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είμαστε όλοι διαιρεμένοι. Και το να φτάσουμε σε κοινή θέση πολύ συχνά οδηγεί σε επιδείνωση αντί για βελτίωση. Γιατί υπάρχει ένας πολτός, ας πούμε, από πράγματα παρά ξεκάθαροι ορισμοί. Στο εσωτερικό επίσης της έκθεσης, δυστυχώς, ως συνήθως, δεν μπήκε μία επίκριση έντονη για την ε, συνταγή αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που απέτυχε και που βασίζεται στην λιτότητα, στις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Τρεις πυλώνες που απέτυχαν, δυστυχώς. Ε, επί χρόνια τώρα αυτή η συνταγή δεν ε, μας εξασφάλισε την ε, έξοδο από την κρίση. Αντίθετα, επιδεινώθηκε κοινωνικός πώς η κρίση και βλέπουμε τι γίνεται στο εκλογικό μέτωπο. Έχουμε ε, το, τους εκλογείς να παραπέουν ε, προς τα άκρα, κυρίως την άκρα δεξιά. αυτές οι ιδεολογικές έτσι, περιπέτειες οφείλονται σε αυτές τις πολιτικές αποτυχημένες που συνεχίζουμε να πιέζουμε, να σπρώχνουμε για να περάσουν. Αντί να κάνουμε μια κριτική και αντί να αλλάξουμε τροχιά στο πλαίσιο της διακυβέρνησης. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που είναι λάθος ε, στην νομισματική ένωση. Δεν υπάρχει καμία κριτική εδώ. Δεν βλέπετε δεν, και δεν αναφέρετε τις ανισορροπίες για την νομισματική ένωση, για το ευρώ, δεν υπάρχει μια κριτική για τις οικονομικές ανισορροπίες που προκλήθηκαν στην νομισματική ένωση. Παραδείγματο χάρη το υπερβολικό πλεόνασμα που έχουν κάποιε χώρε όπω η Γερμανία και η Ολλανδία. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί είναι ανισορροπίε πολύ πιο σοβαρέ σε σχέση με άλλε που αντίθετα εντοπίζονται ξανά και ξανά και στυλιτεύονται αυτός ο ρόλος της Κομισιόν που πάει και τιμωρεί τις ε, αδύναμες χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία ε, αλλά που δεν λέει τίποτα για τις ε, άλλες ανισορροπίες είναι λάθος. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ακριβώς θα πρέπει να τονίσει αυτά τα πράγματα και να τα πει έτσι με τιμιότητα, με ειλικρίνεια, να εντοπίσει το πραγματικό πρόβλημα της ΟΝΕ, που είναι η ανισορροπία λόγω των εμπορικών πλεονασμάτων που έχουν κάποιες χώρες, ενώ κάποιες άλλες χώρες για να γίνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να μειώσουν τους μισθούς, με αποτέλεσμα όλη αυτή την κοινωνική κρίση που σας περιέγραψα στην αρχή της παρέμβασής μου. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να σπρώξει για κάποια αλλαγή. Η ΟΝΕ επίσης είναι μια χαμένη ευκαιρία γιατί την υπερασπίζεστε με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν λέτε ποιο είναι το πρόβλημά τη. Δεν λέτε ποιο είναι το πρόβλημα του ευρώ. Δεν πρόκειται να βγούμε όσο συνεχίζεται με αυτή τη θρησκευτική ευλάβεια από την κρίση του ευρώ. Θα συνεχίζουμε ε, με αυτές τις λύσεις ε, αχταρμά, ας πούμε, μέχρι να διαλυθεί εντελώς με εντελώς ε, άναρχο τρόπο η ευρωζώνη. Εμείς θέλαμε μία διάλυση ε, συντεταγμένη ή ένα πλαίσιο, τόσο ώστε να φτάσουμε σε μία ε, δημοκρατική πραγματική δυνατότητα να βγούμε από την ε, Ευρωζώνη όσες χώρες δεν μπορούν τη στιγμή που οι πολιτικές της Κομισιόν είναι αποτυχημένες. Δεν μπορούμε να έχουμε μία και μόνη νομισματική πολιτική για 19 χώρες που έχουν διαφορετικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, και τα επιτόκια. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Δεν τα δίνει η ΟΝΕ. Δεν τα δίνει η Ευρωζώνη. Όσο συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό το project του ευρώ, δεν μπορούμε να βρίσκουμε συμβιβασμούς ανάμεσα στα τόσο διαφορετικά συμφέροντα που εκφράζονται ε, εκεί μέσα με αυτούς τους αχταρμάδες. Ε, οπότε πολύ λογικό είναι να φτάνουμε σε αυτές τις σε αυτά τα ακροδεξιά ας πούμε και ακραία γενικά ναυάγια, ε, τα οποία θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε όσο συνεχίζουμε. Αυτή είναι η θέση μας και ελπίζω κάποια στιγμή να ξυπνήσει και το Κοινοβούλιο, γιατί οι πολίτες το έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Μπονό, όχι. Πολύ ωραία. Ξανά το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους άλλους συναδέλφους ε, που έχουν βοηθήσει στην ε, κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Άκουσα στην όλη διαδικασία διάφορα επιχειρήματα. Από οικοδομικής πλευράς ε, κάποια από αυτά είναι σεβαστά ε, και άλλα όχι τόσο ίσως αλλά θα επεξεργαστώ την έκθεση δεν θέλω όμως ε, να αρχίζω από την αρχή υπάρχουν ε, κάποιες οριακές συνθήκες που τις οποίες εργαζόμαστε. Στόχος είναι να πάρουμε αυτές τις συνθήκες τις συστάσεις αναχώρα και να βοηθήσουμε με τις υποδείξεις με τις συστάσεις μας να βλέπουμε προς το μέλλον και να τους δώσουμε περισσότερο νόημα. Θεωρώ ότι αν δει κανεί ε, από επενδυτική πλευρά αυτέ τι συστάσει έχουν λογική. Γιατί πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά κάποιο τρόπο σχετίζονται με αυτό το επενδυτικό χάσμα ε, που ανέφερα, αυτό το κενό που δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρωζώνη αλλά και με την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, ιδίως τη ΣΥΠΑ. Αν λοιπόν πούμε ότι είναι ε, στην ε, υποβέλτιστη κατάσταση η ΕΠΑ, μάλλον πάμε λίγο μακριά. Άρα με αυτή τη βάση και με την όθηση που θέλουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις κάθε χρόνο και για τις δημόσιες και για τις ιδιωτικές μιλάω, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε και το βιωτικό επίπεδο, την οικονομική ε, και κοινωνική επίδοση συνολικά της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την ευρύτερη προοπτική προσπαθήσαμε να καταλήξουμε και στις συμβαστικές τροπές που σας παρουσιάσαμε σήμερα. Φυσικά και δεν έχουμε αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη προβλήματα που σχετίζονται με την γέννηση της ε, Ευρωζώνης. Αυτό δεν μας ξεπερνάει, γιατί δεν ήταν στην εντολή μας. Αλλά στην εντολή μας εντάσσεται το να μπορέσουμε να κάνουμε προτάσεις ε, για αλλαγές πολιτικές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση. Είτε είναι βέλτιστη είτε είναι υποβέλτιστη. Αυτός ήταν και ο στόχος και αυτή ήταν ε, και η πρόθεσή μας με τι τροπολογίε που καταθέσαμε. Ευχαριστώ πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς, ζητή τους και όδες. Νομίζω είναι λογικές οι ε, συμβασικές προτάσεις. Και θα τις ψηφίσουμε και σήμερα μάλιστα, το μεσημέρι. Εδώ ολοκληρώνουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ θερμός.